Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω θερμά στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Έχουμε διερμηνία από και προς όλες τις γλώσσες εκτός από τα εσθονικά. Αύριο έχουμε ομάδα επισκεπτών της Μπάρβαρα Βάιλερ ε, σας καλωσορίζουμε και επίσης έχουμε ένα νέο μέλος της Επιτροπής μας που δεν έχω δει ακόμα, την Μαρτίνα Άντερσον, που θα αντικαταστήσει την ε, συνάδελφο Ντεπριούν. Θα την ε, καλωσορίσω όταν ε, έρθει. Τέταρτον, να ανακοινώσω ότι έχουμε κοινή ακρόαση την Τετάρτη από τις 3 και 4 μέχρι τις 5 και 4 το απόγευμα στην αίθουσα Α1G2 στο ASP, στο κτίριο Αλθιέρο Πινέλη, μαζί με τους ε, συναδέλφους από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αλλαγή του κλίματος. Ε, σας προσκαλώ λοιπόν να συμμετάσχετε. και έχουμε μία γραπτή έκθεση ε, σχετικά με την αποστολή στην ε, Λευκοσία της Κύπρου. Υπάρχουν όλα αυτά ε, στην ιστοσελίδα μας. Τρίτη ανακοίνωση, κάτι καινούριο και περιμένω να δω αν θα υπάρξει κάποια αντίρρηση. Τρία μέτρα, 12 εκατοστά και 5 χιλιοστά ε, είχε το ύψος των πρακτικών της συνεδρίασής μας, περισσότερο από πιο ψηλό από έναν άνθρωπο δηλαδή, ε, και γι' αυτό προτείνεται να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά τα πρακτικά. Εάν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση θα υιοθετήσουμε αυτό ε, για να προστατεύσουμε τα δέντρα μας. Ε, ο συνάδελφος Καρλ Χάις Φλόρενς λέει ίσως να χρειαζόμαστε λιγότερα πρακτικά. Επασχεπτώσει τόσα έχουμε. Αναλυτικά λοιπόν ε, καταγράφουμε ε, τι γίνεται στις συνεδριάσεις μας. Και τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω τον, προσκεκλημένο μας, τον σημερινό προσκεκλημένο μας, τον Υπουργό Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σταύρο Μαλά. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας και περιμένουμε αγωνίως να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε για το επόμενο εξάμεινο. Τι μας περιμένει το, το Σαββατοκύριακο. Ε, ε συμμετείχα στην ε, άτυπη συνάντηση των ε, Υπουργών Περιβάλλοντος στην Κύπρο. Ε, ήταν πολύ καλά οργανωμένη η επίσκεψη αυτή. Ε, περιμένω εναγωνίως να δω τι θα μας φέρει η Κυπριακή Προεδρία. Πρώτα θα δώσουμε τον ε, λόγο στον προσκεκλημένο μας ε, και κατόπιν θα έχουμε έναν γύρο ε, με ερωτήσεις από τους συντονιστές και μετά θα πάρουν το λόγο οι άλλοι συνάδελφοί μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε, Υπουργό. κύριε Υπουργέ. Good afternoon, everybody. Dear Chairman. Αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πράγματι είναι μεγάλη τιμή για μένα να μπορώ να απευθύνομαι σε εσά, να είμαι μπροστά σα σήμερα και να παρουσιάζω το πρόγραμμα και του στόχου τη ε, Κυπριακή Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον τομέα τη υγεία. Προσβλέπω σε μια ανοιχτή συζήτηση με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πώς να προωθηθεί ε, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσης στον τομέα αυτό. Η συνθήκη της Λισαβόνας αναμφασβήτητα έχει εισάγει μια πιο ενεργή διαδικασία ευρωπαϊκού κεκτημένου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επεκτείνει τις εξουσίες του ως νομοθετικός φορέας με την προσθήκη περίπου 40 νέων τομέων υπό το πλαίσιο της διαδικασίας συναποφάσεως και έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει σε θέματα που άπτονται του πολιετούς χρηματοπιστωτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Ταυτόχρονα αυτές οι αυξημένες εξουσίες οι οποίες έχουν δοθεί συνεπάγονται μεγαλύτερες ευθύνες προς τους πολίτες, τα εθνικά κοινοβούλια και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κυπριακή Προεδρία καλωσορίζει θερμά αυτές τις αλλαγές και προσβλέπει στην δημιουργία και παγίωση διαδραστικής επικοινωνίας και συνεργασίας με το Κοινοβούλιο σε ένα φάσμα δημόσιων, θεμάτων δημοσίας υγείας που θα βοηθήσουν την υλοποίηση ε, καλύτερης υγείας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Κατά τη διάρκεια του επικειμένου εξαμήνου στοχεύουμε να συνεχίσουμε επί των βασικών προτεραιοτήτων που έχουν καταρτιστεί από την Προεδρία του, του Τρίου στα πλαίσια του προγράμματο αυτό που διαρκεί 18 μήνε και εστιαζόμαστε σε τρει βασικέ γραμμέ δράση. Πρώτα απ' όλα, μη μεταδοτικέ ασθένειε, τονίζοντα την υγιή γύρανση, Δεύτερον, ασθένειες χωρίς σύνορα. Και τρίτον, καινοτομία και ευέλτιστες πρακτικές. Έξι μήνες είναι μια σύντομη περίοδος για να πετύχει κανείς θαύματα, αλλά έχω την πεποίθηση ότι αν συνεργαστούμε σε ένα πνεύμα επικοδομητικού διαλόγου και αμοιβαία κατανόησης, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Επιτρέψτε μου τώρα να ξεκινήσω παρουσιάζοντάς σας το πρόγραμμα και τους στόχους της Προεδρίας μας στον τομέα της υγείας. Το πρόγραμμά μας θα εστιαστεί επί τεσσάρων βασικών αξώνων. Πρώτον, διασυνοριακές απειλές για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, εστιαζόμενοι επί των μεταδοτικών ασθενειών. Δεύτερον, δωρεά οργάνων και μεταμοσχεύσεις. Τρίτον, υγιής γύρανσης καθ, όλη τη διάρκεια του κύκλου της ζωής. Και τέταρτον, καινοτόμε προσεγγίσεις όσον αφορά την περίθαλψη στην υγεία, στον τομέα της υγείας. Η πρώτη προτεραιότητά μας όσον αφορά τις δυσυνοριακές απειλές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικέ χώρες θα εστιαστεί επί των μεταδοτικών ασθενειών. Και αυτό είναι κάτι που προέρχεται από την πρόσφατη εμπειρία από τον H1N1, από τη γρήπη αυτή και την, ε, τις επιδημίες E. coli, που εντόπισαν, έδειξαν ότι χρειάζονται πιο συντονισμένε δράσει, όχι μόνο εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω, αλλά χρειάζεται συντονισμό και με γειτονικέ χώρε. Η σημασία αυτού του τομέα ήδη έχει εντοπιστεί και από την ευρωπαϊκή και τη διεθνή κοινότητα και χρειάζονται, μάλλον έχουν ήδη δρομολογηθεί οι αναγκαίε δράσει προ αυτή την κατεύθυνση. Οι πιο πρόσφατε συζητήσει όσον αφορά την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι διασυνοριακέ απειλέ για την υγεία είναι κάτι που σίγουρα δημιουργεί μια δυνατότητα για ένα νομικό πλαίσιο, τη δημιουργία ενό νομικού πλαισίου σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για αυτό το σκοπό, μια διάσκεψη σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων οργανώθηκε στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα. Η διάσκεψη συνάθρισε διάφορου ε, ενδιαφερομένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι γειτονικέ χώρε τη Ανατολική Μεσογείου και, και ξεκίνησαν σχετικές συζητήσεις όσον αφορά τα σύγχρονα θέματα της δημιουργίας δυναμικού όσον αφορά την πρόληψη, εποπτεία, έγκαιρη προειδοποίηση και αποτελεσματικό έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών. Επίσης, δόθηκε έμφαση στην υπογράμμιση της ανάγκης για συντονισμένες δράσεις μεταξύ των κρατών μερών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των γειτονικών χωρών στους τομείς της προλήψεως και του ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών. Τα συμπεράσματα της διασκέψεως θα υποβληθούν στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας που θα διεξαχθεί στην ε, Λευκοσία αύριο. Η δεύτερη, ο δεύτερος άξονας μας είναι η δωρεά οργάνων και οι μεταμοσχεύσεις. Είναι μια ίστατη πράξη αλτρουισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης που μπορεί να είναι μόνον επωφελής για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που το έχουν ανάγκη λαμβάνοντα υπόψη το μεγάλο αριθμό ασθενών που ωφελούνται από έναν συμβατό δότη, την οικονομική αποτελεσματικότητα της μεταμόσχευσης, καθώς και το μεγάλο αριθμό των ασθενών που είναι σε λίστες αναμονής για συμβατό μόσχευμα, τώρα είναι ανάγκη για περαιτέρω συντονισμένες δράσεις όσον αφορά την αύξηση της ευαισθητοποίησης στο θέμα αυτό. Εργαζόμενοι προς αυτή την κατεύθυνση, η Προεδρία μας θα ετοιμάσει και θα προωθήσει υιοθέτηση αντιστοίχων συμπερασμάτων Συμβουλίου που θα ζητούν περαιτέρω δράση στον τομέα της δωρεάς των οργάνων και της μεταμόσχευσης. Όλος ιδιαίτερος υπό το φως της επικείμενης ενδιάμεσης αξιολόγησης του σχεδίου δράσης για τη δωρεά οργάνων και ε, της μεταμοσχεύσης για την περίοδο 2009-2013. Η τρίτη ο τρίτος άξονας είναι η υγιής γύρανσης ε, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Είναι ένας τομέας που δείχνει τη σημασία που έχει η πρόληψη των ασθενειών και η προώθηση της υγείας σε κάθε στάδιο της ζωής και κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου της ζωής, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται μια υγιής γύρανση. Ιδιαίτερα στα πλαίσια του ισχύοντος του παρόντος οικονομικού πλαισίου και της τάσεως προς γύρανση του πληθυσμού, το να δημιουργηθεί μια διαδικασία για την υγιή γύρανση από τα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί να εξασφαλίσει παραγωγικό πληθυσμό, να ελαχιστοποιήσει τη ζήτηση για περιθάψεις για περίθαλψη που σχετίζεται με χρόνια ασθένειας και συνεπώς θα μειωθεί και το κόστος της περίθαλψης και θα προωθηθεί περισσότερο η ανάπτυξη παραγωγικότητα. Αυτή η προτεραιότητα θα είναι το θέμα των συζητήσεων κατά τη διάρκεια μια διάσκεψη Προεδρία υψηλού επίπεδου με θέμα ε, την υγιή γύρανση κατά διάρκεια του κύκλου ζωή. Αυτή η διάσκεψη έχει σαν στόχο να ε, συναθρήσει ενδιαφερομένου από διάφορου τομεί τη υγεία για να συζητήσουν τα υφιστάμενα στοιχεία και τι βέλτιστε πρακτικέ και συμφωνία για την μελλοντική αντιμετώπιση. Τα αποτελέσματα τη διάσκεψεω θα είναι η βάση για την κατάρτιση συμπερασμάτων του Συμβουλίου για υγιή γύρανση σαν μια συνεχή διαδικασία κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωή, θα εντοπιστούν οι τάσει οι τρέχουσε, θα υπογραμμιστεί η σημασία τη υγεία σαν διατομιακή ε, προσέγγιση και θα ζητηθεί περαιτέρω δράση. Και τέλο, αλλά εξίσου σημαντική προσέγγιση είναι η καινοτόμω προσεγγίση όσον αφορά την περίθαψη στον τομέα τη υγεία. Ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 που συμφωνήθηκε τον Μάρτιο του 2010 που καλεί για μια καινοτόμα ένωση, θεωρούμε ότι το, ένα σύστημα περίθαψης υγείας μπορεί να λειτουργεί σαν οικοσύστημα για ανοιχτή καινοτομία που μπορεί να συνεπιφέρει διάφορους φορείς από διάφορους τομείς και να δημιουργήσει διάφορες συνέργειες. Η παρούσα ε, τάση προς περισσότερη καινοτομία μας υποχρεώνει να δούμε εκτός των συμβατικών εργαλείων που διαθέτουμε. Ανοιχτή καινοτομία ε, είναι μια νέα έννοια που δοκιμάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τη μορφή των, των βάσεων κοινών τεχνολογιών σε ορισμένου τομεί έρευνα. Βασικό μα στόχο είναι να προωθήσουμε την περίθαλψη στον τομέα τη υγεία σε πολυτεμιακό και διατομιακό επίπεδο. Οι εταιρείε που αναπτύσσουν καινοτόμα φάρμακα, οι εταιρείε που ενδιαφέρονται για εφαρμογέ όσον αφορά την πληροφορική στον τομέα τη υγεία, με καινοτόμου τρόπου, οι εταιρείε που κατασκευάζουν τρόφιμα για παιδιά, πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονε όσον αφορά την προσωπική ιατρική, θα είναι από του βασικού συμμετέχοντε σε αυτή τη διάσκεψη που θα λάβει η χώρα στη Λάρνακα τον Οκτώβριο. Επιτρέψτε μου τώρα να κινηθώ προς την παρουσίαση του, των νομοθετικών χαρτοφυλακίων που απαρτίζουν το πρόγραμμα εργασιών της Προεδρίας μας στον τομέα της υγείας. Πριν προχωρήσω στην παρουσίασή μου, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η γενικότερη αρχή που θα διαπνέει την προσέγγισή μας και εντός της ομάδας εργασίας και σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο θα είναι ένα πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού. Όμως θα ήθελα να τονίσω ότι και η αποτελεσματικότητα ή ασδήποτε δράσεις, κυρίως όσον αφορά το πρόγραμμα Υγεία για Ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την οικονομική υποστήριξη. Τα θαύματα δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω ενός προγράμματος με προτινόμενο προπολογισμό 446 εκατομμυρίων ευρώ για μια περίοδο επταετή. Πρώτο χαρτοφυλάκιο, η πρόταση κανονισμού όσον αφορά ε, τη δημιουργία ενός προγράμματος για την, υγεία για την ανάπτυξη στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-2020. Πρόκειται περί ενός μέσου ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή της κοινοτική πολιτικής και των στόχων που έχει θέσει στην υγεία. Συζητήσει στο Συμβούλιο επί Προεδρίας ε, προχώρησαν ε, σε μεγάλο βάθος και υπάρχει μερική συμφωνία επί του θέματος και πετέφθη στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ της 22 Ιουνίου. Η Κυπριακή Προεδρία προσβλέπει σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτω ώστε να πετύχει πλήρη συμφωνία όσον αφορά το περιεχόμενο τη προτάσεω και να υιοθετηθεί το χαρτοφυλάκιο σε μια μερική συμφωνία πρώτη ανάγνωση που εξαρτάται από τη συμφωνία επί του προπολογισμού για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχω υπόψη μου τι μεγάλε τροπολογίε που έχει προτείνει το Κοινοβούλιο και όλο ιδιαίτερο εκείνου που εστιάζονται επί ενδεχόμενων ασυσοτήτων στον τομέα τη υγεία που είναι συνεπαγωγή τη οικονομική κρίση. Πράγματι, συμμερίζομαι αυτές τις ανησυχίες και ελπίζω ότι τα ακόλουθα ετήσια προγράμματα εργασίας θα διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις έκτακτες περιστάσεις που περνούν εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες και θα περάσουν και που έχουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία. Δεύτερο χαρτοφυλάκιο, η πρόταση για μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία. Αυτό είναι πολύ συζητημένο θέμα και σχετίζεται με την προστασία όλων των Ευρωπαίων πολιτών από ένα ευρύ φάσμα απειλών για την υγεία όπως βιολογικές απειλές, χημικές, τέτοιες ή περιβαλλοντικής φύσεως και κάνει προβλέψεις για αποτελεσματικότερο έλεγχο και συντονισμένη ανταπόκριση στην περίπτωση μιας κρίσης. Επίσης ασχολείται με διάφορες βασικές πτυχές της ασφάλειας της υγείας συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας ε, συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωση, εποπτεία και ανταπόκρισης όσον αφορά τι απειλέ, όπω αυτέ που ε, δημιουργούνται από τις ε, μεταδοτικέ ασθένειε. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων που ξεκίνησαν στον, ε, στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου από την προηγούμενη Προεδρία επιτρέπουν στην Κυπριακή Προεδρία να προχωρήσει περαιτέρω στο χαρτοφυλάκι αυτό και να συζητήσει και να διαπραγματευτεί περαιτέρω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπω ότι οι μακροσκελείς συζητήσεις θα λάβουν χώρα και εντός του Συμβουλίου και μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να αναλάβουμε αυτό το καθήκον με θετικότατο τρόπο, λαμβάνοντα υπόψη αυτά που συνέβησαν στο παρελθόν, με, όταν σοβαρέ επιδημίε ανησύχησαν την Ευρώπη και θα εξασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε θα αποφασίσουμε πλήρως και αποτελεσματικά θα εξυπηρετεί το σκοπό καλύτερης και πια ομοιόμορφης δράσης σε όλη την Ευρώπη. Ο τρίτο τομέα, το τρίτο χαρτοφυλάκιο, αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα και είναι η πρόταση για την αναθεώρηση τη οδηγία 2001 κάθετο 20 ε, Ευρωπαϊκή ε, ΕΟΚ για κλινικέ δοκιμέ. Σχετίζεται με την αναθεώρηση των απαιτήσεων για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών επί ανθρώπων και έχει σαν στόχο την ανακάλυψη ή επαλήθευση δράσεων Ενό ή περισσότερων ιατρικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων και έχουμε σαν στόχο την εναρμόνιση της αξιολόγησης και της αδειοδότηση ε, των κλινικών δοκιμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει μια πρόταση για κανονισμό κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και περιμένουμε να προωθήσουμε αυτό το χαρτοφυλάκιο και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία όσον αφορά το πλαίσιο αυτό σε επίπεδο Συμβουλίου. Τέταρτο χαρτοφυλάκιο, η πρόταση οδηγία 89 κάθετο 105 ΕΟΚ, που σχετίζεται με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων για την ανθρώπινη χρήση και τη συμπερίληψή του στο πεδίο εφαρμογή των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων. Αυτό έχει σαν στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την εγκατάσταση τη οδηγία 89 κάθετο 105 ΕΟΚ. Η προηγούμενη οδηγία θεωρείται ότι δεν αντικατοπτρίζει πλέον τον περίπλοκο χαρακτήρα της τιμολόγησης και των διαδικασιών επιστροφής των χρημάτων εντός των κρατών μελών. Η νέα οδηγία επουδενή δεν επηρεάζει τις εθνικές πολιτικές που σχετίζονται με την τιμολόγηση και τη διοργάνωση των κοινωνικών ασφαλιστικών συστημάτων, εκτός στο βαθμό που θεωρείται αυτός αναγκαίος για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια. Η συζήτηση της πρότασης σε επίπεδο ομάδας εργασίας όσον αφορά τα φαρμακευτικά και τις ιατρικές συσκευές ξεκίνησε από την Δανέζικη Προεδρία και θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της δικής μας Προεδρίας. Το ε, έργο αυτό θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου εκεί ξανά στενή συνεργασία απαιτείται και μια συζήτηση προσανατολισμού θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ το Δεκέμβριο 2012. Πέμπτο χαρτοφυλάκιο, η αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου όσον αφορά τις ιατρικές συσκευέ που απαρτίζεται από την αναθεώρηση των προτάσεων για οδηγία όσον αφορά τις ιατρικές συσκευέ και αναστολή της εφαρμογής οδηγίας 90-85 και 93-42 και της πρότασης οδηγίας που αφορά την in vitro διαγνωστικές συσκευές και αναστολή ισχύω της οδηγίας 9879 που έχει σαν στόχο την προστασία της υγεία και της ασφάλειας των πολιτών τη ευρωπαϊκή Ενώσεω και την εξασφάλιση της ευρύθμου λειτουργίας ενία αγορά. Τα πρόσφατα γεγονότα με τα εμφυτεύματα στήθου και τα, και τα υποκατάστατα όσον αφορά ε, τη, διάφορες, ε, διάφορες αθρώσεις αποκάλυψαν την ανάγκη για αυξημένο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών για να υπάρχει ασφάλεια. Η Προεδρία μα θα ξεκινήσει τι συζητήσει στο Συμβούλιο και την ομάδα εργασία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαπραγματευτούμε την μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή από τα κράτη-μέλη εντό του προβλεπωμένου χρονοδιαγράμματο. Εξή, το κόπο να αναφέρουμε ότι στόχο μα είναι να συνεχίσουμε την εργασία μα όσον αφορά την εφαρμογή του φεσταμένου σχεδίου δράση, όσον αφορά τι ιατρικέ συσκευέ, για να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία των φορέων κοινοποίησεω, το συντονισμό, ε, συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ 100 μελών και την ανιχνευσιμότητα, ώστε να εγγυόμεθα την ασφάλεια των ασθενών στα πλαίσια των συζητήσεων για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου. Έκτο χαρτοφυλάκιο πρόταση για κανονισμό όσον αφορά τα τρόφιμα για τα παιδιά, τα νέα παιδιά και τα βρέφη και τα τρόφιμα για ειδικέ ιατρικού σκοπού και θέλουμε να διευκρινίσουμε, να πλουστεύσουμε το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα τρόφιμα που έχουν ιδιαίτερε διατροφικέ χρήσει. Η Κυπριακή Προεδρία θα προσπαθήσει να βρει ε, το μέσο όρο όσον αφορά τι διαφορέ που υπάρχουν μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση του χαρτοφυλακίου ε, και ελπίζουμε αυτό να γίνει σε ένα πρώιμο, σε ένα αρχικό στάδιο τη δεύτερη ανάγνωση. Μετά έχουμε μια πρόταση όσον αφορά την οδηγία για ε, το πρωινό ε, που έχει σαν στόχο να γραμμίσει τις εξουσίες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη διαχωρισμό μεταξύ κατεξοδότηση πράξεων και εφαρμοστικών πράξεων που δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των άρθρων 290 και 291 τη συνθήκη όσον αφορά τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και να δοθούν περαιτέρω κατεξοδότηση εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Δανική Προεδρία ξεκίνησε συζητήσει στο Συμβούλιο και η Κυπριακή Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια τόσο ώστε να προχωρήσει ή και να ολοκληρωθεί η συζήτηση επί του χαρτοφυλακίου αυτού. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αυτή, αυτό εν γέννη ήταν το πρόγραμμά μας για την υγεία και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Έχουμε επίγνωση του καθήκοντος που μας περιμένει, του έργου που μας περιμένει και των ευαισθησιών ε, που αφορούν διάφορα θέματα. Όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και λύση και βασιζόμαστε κατά πολύ στην εργασία μας με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο και μπορούμε και θα έπρεπε να προχωρήσουμε όσον αφορά θέματα πολιτικής υγείας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Συζητώντας τα θέματα που υπογραμμίστηκαν προηγουμένως, κανείς δεν μπορεί να λησμονήσει ποιο είναι το γενικό περιβάλλον που επικρατεί σε όλη την Ευρώπη. Η οικονομική κρίση οδηγεί σε δημογραφικές αλλαγές και ασκεί σοβαρές πιέσεις επί των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης όλων των κρατών μελών. Εν τη ελήψη λοιπόν οικονομικών πόρων, αυτή είναι η στιγμή να είμαστε δημιουργικοί. Τα γεγονότα εκτελήσονται γύρω μας καθημερινά και συγκλονίζουν τον κοινωνικό και οικονομικό εστό της Ευρώπης με έναν τρόπο ανευπροηγουμένο. Πράγματι μπορεί να πει κανείς ότι η Ευρώπη έφτασε περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, την πιο δύσκολη περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως, όπως στην εποχή του πολέμου η αλληλεγγύη είναι μια φυσική ανθρώπινη αντίδραση προσπαθώντας να επιβιώσουν οι άνθρωποι, σε στιγμές ειρήνης η αντίδραση δεν θα έπρεπε να είναι διαφορετική. Ελπίζω ότι όλοι θα ανταποκριθούμε στις περιστάσεις και θα δείξουμε την ευρωπαϊκή ελληνική που όλοι ε, ρητορικά ε, εγκρίνουμε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους τέσσερις συζητητές. Ήταν πολύ καλή συζήτηση που διεξήχθη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Κυπριακής Προεδρίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την ε, εξαιρετική επισκόπηση που μας παρουσιάσατε των επόμενων έξι μηνών. Πολλά θέματα έχετε στο θεματολόγιο σας. Βλέπω τα χέρια που σηκώνονται. Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο γύρο ε, θα ακούσουμε του ε, συντονιστέ. Ε, Συντονιστή τη ομάδα του ΕΛΚ είναι ο Πέτερ Λίζε. Παρακαλώ, Πέτερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Προεδρεύοντα. Τρία θέματα πολύ σύντομα. Επικροτώ το γεγονό ότι θέλετε να αντιμετωπίσετε τα βασικά ζητήματα στην κατά τη διάρκεια τη Προεδρία σα, ιδιαίτερα το θέμα των δωρητών οργάνων. Είναι κάτι που μα ενδιαφέρει πολύ εδώ. Πολλοί άνθρωποι περιμένουν να λάβουν κάποιο όργανο. Δεν έχουμε πετύχει αρκετά εδώ στην Ευρώπη. Θα ήθελα να επιστήσω την ε, προσοχή σας σε ένα αίτημα του Κοινοβουλίου να καταπολεμήσουμε το εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων. Την προηγούμενη εβδομάδα ε, επικοινώνησε μαζί μου το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο ε, που εργάζεται πάνω σε ένα πρωτόκολλο για αντιμετώπιση του εμπορίου ανθρωπίνων οργάνων ε, δεν ε, εκπροσωπείται εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν χρήσιμο να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, σύντομα για δύο νομοθετικά θέματα. Το σχέδιο δράσης για την υγεία. Έχει λάβει νέο τίτλο από την Επιτροπή μας. Θέλουμε να λέγεται Health for Growth and Citizens, ώστε να αναφέρονται και οι ε, πολίτες, να μην, δίνουν, να μην δίνουμε την εντύπωση ότι ε, το θέμα αυτό έχει να κάνει μόνο με την οικονομία, όσο σημαντική και αν είναι ε, η οικονομία σε εποχές κρίσης. Ε, πρέπει δηλαδή να είναι σαφές ότι μας ενδιαφέρει η, η υγεία των πολιτών. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη διαμηνία, τώρα διορθώθηκε ωραία υπήρχε διερμηνία προ τα αγγλικά. Παρακαλώ. Ε, η τελευταία μου παρατήρηση, συνεχίζει ο κ. Λίζε, να σας ευχαριστήσω που αναφερθήκατε στο θέμα των κλινικών δοκιμών. Ελπίζω κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας σας να υπάρξει σχετική πρόταση από την Επιτροπή πριν το καλοκαίρι. Ε, πρέπει Ε, να κάνουμε κάτι επειδή ε, επιστήμονες ε, που θέλουν να κάνουν δοκιμές δυσκολεύονται λόγω της υπάρχουσας οδηγίας. Το Κοινοβούλιο έχει υποδείξει τα προβλήματα ήδη πριν 10 χρόνια όταν διαπραγματευτήκαμε την οδηγία πρέπει να πείσουμε το Συμβούλιο ότι χρειαζόμαστε ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία προς όφελος των ασθενών ε, ε, του, του, σχετικού τομέα και ε, και των δοκιμών. Ευχαριστώ πολύ, Ιντάγμα Ροτ Πέρεντ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, Λίντα. Ευχαριστώ, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για τις φιλοδοξίες σας. Μερικές φορές λέμε ότι λες εσμό, ότι καλύτερα να έχουμε κάτι λιγότερο. Είμαι όμως αισιόδοξη ότι θα πετύχετε. Ε, αν ήμουν στη θέση σας ε, και αν μπορούσα να σας ε, δώσω μια συμβουλή, θα βασιζόμουν περισσότερο στη, στο νομοθετικό και λιγότερο στο μη νομοθετικό κομμάτι της δουλειάς. μιλάτε για διασυνοριακές απειλές προς την υγεία και αναζητάτε ένα νομικό πλαίσιο. Σκεφτείτε τι έγινε με την ε, νομοθεσία μας για τη διασυνοριακή ε, γιατρική περίθαλψη ε, και πόσο φιλόδοξα ήταν τα κράτη-μέλη. Αν ήσασταν ήδη υπουργό, τότε μπορεί να το θυμάστε. θα, ήθελα πάντως να σας συγχαρώ, όπως ανέφερε και ο κύριος Λίζε. Θα ήθελα να επανέλθω σε δύο παρατηρήσεις. Ε, δεν θα αναφερθώ ε, στην ε, σχετική οδηγία, διότι η συνάδελφοι θα αναφέρει σε αυτό, αλλά όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές, αναφέρθηκε ο Πέτερ Λίζε στο θέμα αυτό. Ελπίζω τα κράτη-μέλη να πρέπει να μοιραστούν δεδομένα και εμπειρογνωμοσύνη ώστε να συγκεντρώνεται η ε, αριστεία ε, και τα δεδομένα, να μην ε, έχουμε ο καθένα το μικρό του βασίλειο, να γνωρίζουμε ότι οι κλινικέ δοκιμέ είναι ένα νόμισμα με δύο πλευρέ. Θα πρέπει αφενό να προστατεύσουμε αυτού που συμμετέχουν στι κλινικέ δοκιμέ, από την άλλη θα πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία. Και φτάνω στι ιατρικέ συσκευέ και αυτό με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Κάπω ανατρίχιασα όταν μου είπατε ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε την λειτουργία των φορέων κοινοποίηση. Ελπίζω να μην προδικάζεται όχι μόνο το περιεχόμενο της νομοθεσίας, αλλά και το περιεχόμενο των συζητήσεων εδώ, διότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η μοίρα των φορέων κοινοποίηση. Ε, χρειαζόμαστε τέτοιου φορεί και αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση προ εσά. Ε, όσον αφορά τα διάφορα γιατρικά βοηθήματα, πιστεύετε ότι όλα θα πρέπει να, ε, ε να περνάνε από κάποια αρχή κοινοποίηση ή πιστεύετε ότι κάποια πρέπει να λαμβάνουν άδεια, να πιστοποιούνται. Εάν ε, χρειάζεται μία άδεια, ε, για παράδειγμα, εάν έχουμε να κάνουμε με ένα βοήθημα που αποτελεί εργαλείο για μια δραστική ουσία ή εάν ε, το ίδιο περιέχει μια δραστική ουσία. Δεν πιστεύετε ότι σε αυτές τι περιπτώσεις χρειάζεται άδεια, για παράδειγμα, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ή από κάποιον εθνικό οργανισμό. Και ταυτόχρονα πιστεύω ότι γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πριν από οποιοδήποτε ε, σκάνδαλο για τα εμφυτεύματα στήθους μα οδήγησαν σε αναθεώρηση της νομοθεσίας ε, το Κοινοβούλιο ήθελε κάτι τέτοιο, είχαμε σχετική έκθεση. Συμφωνείτε μαζί μου ότι όσον αφορά τα ιατρικά βοηθήματα θα πρέπει να είμαστε πολύ ε, σαφείς ε, να έχουμε διάφορες κατηγορίες, να έχουμε αρχή κοινοποίηση για, για τα πιο απλά γιατρικά βοηθήματα, να υπάρχει ένα, ένας φορέας καταχώρηση σε κάθε κράτος μέλος και να, να συνεννοούνται μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και για τους παραγωγούς ε, των ε, των ιατρικών βοηθημάτων. Η Γερμανία έχει 18 φορείς κοινοποίησης και ο κάθε παραγωγός μπορεί να επιλέξει που θα ε, υποβάλει το προϊόν, το, το του και γι' αυτό άλλωστε ο παραγωγός αυτών των αμφιλεγόμενων εμφυτευμάτων ε, στήθου ε, επέλεξε στην Γερμανία να κάνει την καταχώρηση. Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι εφόσον περιμένουμε από την ε, Κομισιόν να υποβάλει πρόταση για τις κλινικές δοκιμές πριν το καλοκαίρι και για τα ιατρικά βοηθήματα το Σεπτέμβριο, μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι θα σημειώσετε πρόοδο κατά διάρκεια της Προεδρίας σας. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Πανάκοβα ε, για τους φιλελεύθερους. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για την παρουσίασή σας. Από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ δύσκολο να διεκπαιρεώσετε τα καθήκοντά σας, διότι από τη μία πλευρά ποτέ καμία προεδρία δεν ε, διέπεται από υπερβολικά μεγάλες φιλοδοξίες για την προώθηση νομοθεσίας για τα θέματα της υγείας, πόσο μάλλον για νομοθεσία η οποία αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένη, και από την άλλη διότι ασκείται, ασκείται πίεση από τις χώρες που ενδιαφέρονται ιδιαίτερως για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και περικοπές. Θα συζητήσετε με τους συναδέλφους σας το μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των περικοπών στον τομέα της υγείας. Είναι αυτό στις προθέσεις σας και μάλιστα αναφέρομαι σε εκείνους ε, που ε, προέρχονται από χώρες όπου ανοιχνεύεται μακροπρόθεσμος αρνητικός αντίκτυπος. Επιπροσθέτως, ως προς την οδηγία για τη διαφάνεια και για τα φαρμακευτικά προϊόντα, θα γνωρίζετε φαντάζομαι τις αρχικές αντιδράσεις των κρατών μελών σε σχέση με το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να μας πείτε την απόψή σας, πώς θα προχωρήσει η πρόταση αυτή, ποιες είναι οι προθέσεις σας. Ποια είναι η κύρια βάση πάνω στην οποία ε, μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής, η κυρία Μαρίνα Γιανακουδάκη από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για μια πολύ συνεκτική παρουσίαση, την οποία καλωσορίζει ιδιαίτερως η δική μου πολιτική ομάδα. Μου άρεσαν ιδιαίτερως τα εξής σχόλια. Εναπουσία οικονομικών πόρων. Ε, στα ελληνικά αυτό θα το σχολίαζα με τον όρο σαφώς. Δεν ξέρω αν είναι σωστό στα ελληνικά, αλλά Πράγματι έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, ως προς το διασωνεωριακό, ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη των Λοιμόξεων και ως προς τις δωρεές. Είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερος, γιατί μόλις ε, δούλεψα πάνω σε μια έκθεση για το θέμα αυτό. Συμφωνώ με αυτά που μας είπε ο Πίτερ. Θα ήθελα όμως να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον εθελούσιο χαρακτήρα και στη μία χρηματική ανταλλαγή. Σίγουρα εργάζεστε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Και τέλος, η γύρανση σε συνθήκες υγείας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και για λόγους υγείας, αλλά και για λόγους οικονομικούς. Όσο πιο υγιής είναι ο πληθυσμός, τόσο λιγότερο στοιχίζει στα κράτη. Σίγουρα είναι κάτι που εξετάζεται. Σε γενικές γραμμές πρέπει να σας πω ότι εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το πρόγραμμά σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Τελευταίος ομιλητής από πλευράς της ΚΟΕ, η κυρία Σούζα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σημαντική η παρουσίασή σας Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που την ακούσαμε και που μπορέσαμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. Ωστόσο, έχω δύο πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα να απευθύνω και ίσως προκύψουν και αργότερα κάποια άλλα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Πρώτον, ο ορίζοντας 2020. Έχουμε ένα προπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ για 6 χρόνια, 31,7 εκατομμύρια ευρώ για τις πολύ σημαντικές προκλήσεις για την υγεία, για την αηφόρο γεωργία και το καθεξής. Στην πράξη όμως αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε 5,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ένα μικρό σχετικά ποσό, εάν το συγκρίνουμε με το γενικότερο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ε, την οικονομική κρίση που σοβεί στις διάφορες χώρες μέλη, τι πιστεύετε για το ποσό αυτό, θα είναι επαρκές? θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ως προς την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων με αυτά τα χρήματα. Αυτό ήταν το πρώτο μου ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα που έχει σχέση με το πρώτο. Μπορείτε λίγο να μας αναπτύξετε το θέμα των ανισοτήτων ως προς την υγεία και των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν στην υγεία. Αυτή τη στιγμή διανύουμε μια περίοδο μεγάλης κρίσης και διαπιστώνουμε ισχυρές ανισότητες όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και στο εσωτερικό διαφόρων κρατών μελών. Τελικά δεν γεφυρώνουμε το χάσμα των ανισοτήτων στην Ευρώπη και τα περισσότερα μέτρα που έχουν ληφθεί πρόσφατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ουσιαστικά κάνουν το χάσμα αυτό ακόμα πιο αγεφύρωτο. Μπορείτε να μας σχολιάσετε με πιο συγκεκριμένο τρόπο τα μέτρα αυτά για την καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Φτάνουμε ε, στο τέλος του πρώτου γύρου ερωτήσεων από πλευρά συντονιστών. Να δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του δύο λεπτά για να απαντήσει τα ερωτήματα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Κύριε Λίζη, βεβαίως, έχουμε επιλέξει ε, τις βασικές πτυχές της ε, δωρεάς οργάνων. Η κινητοποίηση της κοινωνίας και ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει αυτό στην δωρεά οργάνων. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ίσως δεν θα το γνωρίζετε, αλλά μπορώ να σας πω κύριε Λίζε ότι το 1 τρίτο του πληθυσμού της Κύπρου αυτή τη στιγμή είναι δωρητές ε, μυελού των οστών. Έχουμε κινητοποιήσει την ε, κοινωνία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να έχουμε μια πολύ μεγάλη δεξαμενή ανθρώπων, οι οποίοι είναι δωρητές. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο την την κοινωνία και να φανεί ξεκάθαρο ότι με την κινητοποίηση της κοινωνίας μπορούμε να πετύχουμε αυτό το οποίο επιθυμούμε. Ωστόσο βεβαίως και υπάρχει μεγάλη ανάγκη μεταμόσχευσης οργάνων. Ε, είναι ένα, ε, ε, έχει οικονομική διάσταση το θέμα αυτό, αλλά έχει και κοινωνική διάσταση. Σε μεγάλο βαθμό χρειάζεται περισσότερο συντονισμός, περισσότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε να διευρύνουμε αυτή τη συνεργασία, θέλουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ώστε να υπάρχει όσο δυνατόν πιο ευρεία πρόσβαση σε όργανα σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, ως προς το θέμα του τράφικιν, και το λέω και ως ε, Υπουργός Υγείας, Πράγματι, έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου λόγω αναποτελεσματικής νομοθεσίας έχει ανοίξει παράθυρο για την εμπορία οργάνων και όχι για την δωρεά οργάνων. Είναι κάτι που συμβαίνει στην Ευρώπη, πρέπει να το ε, ε, ε, πούμε και να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας. Θεωρώ ότι μια πιο ομοιόμορφη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών πραγματικά ε, θα προστατεύσει όλους μας από την εμπορία οργάνων και θα φράξει το δρόμο ε, σε αυτούς που την ε, προσδοκούν. Τώρα, έχει γίνει πολλή συζήτηση για το όνομα «Υγεία για την Ανάπτυξη». Health for Growth. Αυτό είναι που προτείνει το Κοινοβούλιο για τους πολίτες. Δεν ξέρουμε τελικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ποια θα είναι η τελική έκβαση των συζητήσεων. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής. Το βεληνικές αυτού του προγράμματος δεν είναι τεράστιο. Μιλούμε για 446 εκατομμύρια ευρώ ε, σε ένα βάθος χρόνου 6 ή 7 ετών. Επομένως, ε, με τις ε, συγκεκριμένες παρεμβάσεις, η διαφορά τελικά που θα σημειωθεί με αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να το πούμε ειλικρινά, δεν θα είναι και τόσο σπουδαία ή τόσο μεγάλη πια. Όπως και να το πούμε τελικά, η ουσία του θέματος το οικονομικό διατάφτα είναι αυτό που θα κάνει και τη διαφορά. Τώρα, ε, για τις κλινικές δοκιμές. Είναι κάτι που υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια. Να πω το εξής. Γιατί χρειαζόμαστε οδηγία εναρμόνισης κλινικών δοκιμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει ουσιαστικό έλλειμμα καινοτόμων φαρμάκων στο μέλλον. Και γιατί θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Διότι η ανακάλυψη αυτών των φαρμάκων αυτή τη στιγμή επιβραδύνεται με πάρα πολύ ε, έντονο ρυθμό. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιβαράδυνση. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, καθυστερεί η ανακάλυψη νέων φαρμάκων είναι οι κλινικές δοκιμές οι οποίες ευθύνονται για το 50% του κόστους για την ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου. Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι λόγοι βεβαίως, τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε, που έχουν να κάνουν με την έρευνα, σε κάποια άλλη ευκαιρία. Επομένως, είναι κάτι που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη τις εναρμονισμένες κλινικές δοκιμές. Όχι μόνο για να έχουμε καινοτόμα φάρμακα, αλλά τα χρειαζόμαστε και για οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να είμαστε σε θέση να δοκιμάζουμε αυτά τα φάρμακα και να έχουμε αποτελέσματα. Υπάρχει δηλαδή και μια οικονομική συνιστόσα εκεί, στις εναρμονισμένες κλινικές δοκιμές. Στρέφομαι τώρα προς την κυρία Ροτμπέρεντ και να σας πω ότι σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Δεν είναι κακό να είναι κανείς φιλόδοξος. Θα είμαστε φιλόδοξοι και με ό,τι καταφέρουμε θα είμαστε μετά ικανοποιημένοι. Τώρα, ως προς την νομοθεσία για τις απειλές ε, της υγείας, συμφωνώ μαζί σας, έχει βαλτώσει κάπως η κατάσταση. Σε επίπεδο Συμβουλίου, όμως, έχουν σημειωθεί κάποιες ε, θεμελιώδεις αλλαγές ε, σε σχέση με την οδηγία αυτή και βλέπω ότι ε, υπάρχει και μία αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη βασική αρχή πίσω από όλα αυτά, η οποία είναι η εξή. Μας χρειάζεται το μέγιστο δυνατό επίπεδο συντονισμού στην Ευρώπη. Γνωρίζετε ότι στο παρελθόν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο και θα έπρεπε να το έχουμε και πρέπει να το αποκτήσουμε. Με το συντονισμό αυτό αποφεύγουμε την ε, δημιουργία καινού χώρου, τελικά να ε, εμφανιστούμε ένα δυναμία υποβολής ε, γνωμοδότησης και άποψης τελικά και έτσι ανοίγουμε το δρόμο ε, οι ιδιώτες να έρχονται και να καλύπτουν το κενό. Το είδαμε αυτό και με τα εμβόλια στο παρελθόν. Αυτή λοιπόν είναι η βασική αρχή και θα κάνουμε το παν να πετύχουμε συμφωνία τουλάχιστον σε επίπεδο Συμβουλίου. Σημειώνω όμως αυτό που μου είπατε ότι πράγματι είναι αυτό εξαιρετικό, εξαιρετικά φιλόδοξο. Αλλά πάντοτε πρέπει να είναι κανείς φιλόδοξος πολύ για να πετύχει έστω και λίγα. Τώρα για τις ιατρικές συσκευές και τα... Ε, ε όλα αυτά τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα. Έχουμε τα, βεβαίως το σκάνδαλο με τα εμφυτεύματα, το γνωστό, τα λαμβάνουμε αυτά, όλα αυτά υπόψη μας, είδαμε ότι κάποιες εθνικές ε, αρχές αρμόδιες υιοθέτησαν διαφορετική άποψη από κάποιες άλλες και τελικά στο Συμβούλιο ε, ήταν εξαιρετικά δύσκολη η παρουσίαση μιας ε, κοινή δήλωσης. Συμφωνήσαμε όμως στο εξής. Ο αρμόδιος επίτροπος για την υγεία εξέδωσε μια δήλωση στην οποία καλεί τα κρατη να καταρτήσουν ένα μητρό, ένα εθνικό μητρό, όπου μπορούμε να εντοπίζουμε ε, οποιονδήποτε πολίτη, ο οποίος, η οποία μάλλον ε, ε, χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα εμφυτεμάτων ε, στήθους. Αυτό είναι μια αρχή και θα είναι και μια βάση για τη συζήτηση της ε, καινούργιας οδηγίας. Δεν έχουμε ακόμα τη νέα πρόταση, αλλά θεωρώ ότι θα ε, περιλαμβάνει μέτρα για το διορισμό και την εποπτεία των ε, φορέων κοινοποίηση και για τον έλεγχο. Σημειώνω αυτό που λέτε και συμφωνώ. Οι φορείς ε, κοινοποίησης αναλαμβάνουν πολύ μεγάλες ευθύνες και μάλιστα ε, για εμφυτεύματα τα οποία έχουν και φαρμακευτικό χαρακτήρα και για τα οποία χρειάζεται ειδική άδεια. Είναι δύσκολο κανείς να χαράξει τα όρια. Αυτό το αποδέχομαι πλήρως και συμφωνώ. Ωστόσο πρέπει να ξεκινήσουμε. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Τώρα, ε, ως προς τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Έχουμε εμπειρία στην Κύπρο για το θέμα αυτό. Αναφερθήκατε στην οικονομική κρίση. Καταρχάς, να πω ότι αυτό που παρατηρώ και που έχω παρατηρήσει είναι ότι η φαρμακοβιομηχανία είναι έτοιμη σε τόσο δύσκολους καιρούς σήμερα να κάνει υποχωρήσεις ως προς τα συστήματα υγείας των κρατών. Αυτό ισχύει, μου το έχουν πει οι ίδιες οι εταιρείε της φαρμακοβιομηχανίας στη δική μας χώρα, αλλά και αλλού. Και εμείς στη δική μας χώρα έχουμε λάβει διάφορα μέτρα για να μειώσουμε το κόστος. Και μάλιστα ε, ήταν και αρκετά αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά. Βεβαίως πρέπει να συζητήσουμε ορισμένα θέματα όπως είναι ο χρόνος και η χρονική συγκυρία διοδότησης ε, για τα καινοτόμα φάρμακα μεταξύ άλλων. Όμως, ως προς την οδηγία αυτή ε, νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό το περιεχόμενο και αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι έχει καταλάβει η φαρμακοβιομηχανία ότι πρέπει να έχει πιο εφικτές τιμές ε, όταν κοστολογεί τα φαρμακά της. Και δεν μας χρειάζεται απαραίτητο μια οδηγία για να το πετύχουμε αυτό. Μπορούμε να τα συζητήσουμε και με άλλους τρόπους. Στρέφομαι τώρα προς την κυρία Γιανακουδάκη για να την ευχαριστήσω καταρχάς για τα θερμά της σχόλια. Την περασμένη εβδομάδα συναντηθήκαμε με τον εκπροσώπους του Οργανισμού για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των ε, Ασθενειών. Και θα ήθελα να πω ότι ο ρόλος που διαδραματίζει αυτός ο οργανισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός για μικρές χώρες όπως είναι η Κύπρος. Και το λέω αυτό διότι οι μικρές χώρες δεν έχουν πάντοτε την απαραίτητη εμπειρία ή εμπειρογνωμοσύνη ή τις απαραίτητες δυνατότητες για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους κρίσεις. Και γι' αυτό στρέφονται προς αυτόν τον οργανισμό ο οποίος παρέχει τις ειδικέ πληροφορίες, ο οποίο έχει ε, πολύ μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία. Είναι κάτι που συνέβη στην περίπτωση του ΙΤΑ 1 1. Τώρα, ως προς τον εθελοντικό χαρακτήρα, να σας πω ότι βεβαίως η κινητοποίηση της κοινωνίας στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως είναι θεμελιώδης και συμφωνούμε απολύτες. Ως προς την ε, γύρενση με υγεία, ε, το healthy aging, αυτό όντως είναι οξύμορο. Ε, φαίνεται οξύμερο, οξύμορο εκ πρώτης όψης. Ωστόσο, η γύρανση με υγεία είναι το αποτέλεσμα διαφόρων βιολογικών διαδικασιών οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα πρώτα στάδια της ζωής ή αργότερα και τελικά, παρόλο που φαίνεται οξύμορος αυτός ο χαρακτηρισμός, έχει πολύ μεγάλο νόημα. Στη συνάντηση υψηλού επίπεδου θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι να γίνονται παρεμβάσεις έγκαιρα, από νωρί στη ζωή. Να, έχ, να εδραιώσουμε υγιείς διατροφικές συνήθειες στα παιδιά, για παράδειγμα. Να αντιμετωπίσουμε τις βασικές αιτίες που ευθύνονται για τα καρδιακιακά νοσήματα και για τον διαβήτη, που είναι οι δύο βασικές κατηγορίες νοσημάτων που επιβαρύνουν τόσο πολύ τα κρατικά, τα εθνικά συστήματα υγείας. Και θέλουμε και να δώσουμε έμφαση στα θέματα που απασχολούν την τρίτη ηλικία. δεν θα περιοριστούμε ε, στις ασθένειες που ταλανίζουν την τρίτη ηλικία, αλλά θα ε, οργανώσουμε και μια προκλητική, αν θέλετε, συζήτηση για τα απορίσματα και τα αποτελέσματα των ερευνών ε, που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για τα βλαστοκύτταρα και τη χρήση αυτών για, σκοπ... για... για θεραπευτικούς σκοπούς. Άλλωστε, αυτά είναι και τα επιχειρήματα των ερευνητών, ότι διεξάγουν έρευνα στα βλαστοκύτταρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ασθένειες της τρίτης ηλικίας. Με αυτή τη συζήτηση λοιπόν θέλουμε να ε, παρουσιάσουμε στους Υπουργούς Υγείας και στους υψηλούς αξιωματούχους τη θέση μας για τα ε, βλαστοκύτταρα, διότι πραγματικά είναι μια σφίζουσα περίοδος ε, αυτή που διανύουν οι ερευνητές βλαστοκυτάρων και πρέπει να γνωρίζουμε τα αποτελέσματά τους. Μπορώ να απαντήσω στο τελευταίο σας ερώτημα σε σχέση με την έρευνα, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, γιατί θα ήθελα πρώτα να ενημερώσω τους αρμόδιους βουλευτές από την Επιτροπή Ήτρε. Σε αυτό το στάδιο μπορώ μόνο να πω ότι είναι ένα πρόγραμμα 80 δις. Και το, το Κοινοβούλιο για πρώτη φορά θέλει αυτό το ποσό να το πάει στα 100 δις και είναι πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο κάνει μια τέτοια παρέμβαση. Ως προς το, την κατανομή αυτού του προϋπολογισμού ε, σας ζητώ συγγνώμη αλλά είναι κάτι που πρέπει να συζητήσω με, τους, ε, με τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε για να μην υπάρξει σύγχυση περί ε, διαφόρων φακέλων. Παρόλο που πραγματικά δύσκολα αντιστέκομαι στον πειρασμό να το συζητήσω το θέμα αυτό με εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για τις ε, συγκεκριμένες και αναλυτικές απαντήσεις ε, που μας δώσατε στις ερωτήσεις των ε, συντονιστών και συναδέρφων. Ξεκινάμε τον ε, δεύτερο γύρο. Άντρες Περέλο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Υπουργό για τις παρουσιάσεις του. Όμως θέλω ένα στοιχείο να μοιραστώ μαζί σας και μία ερώτηση να σας θέσω. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με την κυρία Γιανακουδάκη όταν ε, συντάσαμε το κείμενο για τα εμφυτεύματα. Αυτή τη στιγμή και για τις ε, μεταμοσχεύσεις κυρίως. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, διανύουμε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση και με αυτή την αφορμή γίνονται πάρα πολλές περικοπές παντού. Πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη ε, μιλούν για την ανάγκη να υπάρχει οικονομικό κίνητρο για τις δωρεές οργάνων και για τις μεταμοσχεύσεις. Εγώ διαφωνώ καθέτως και νομίζω ότι πρέπει να ε, πατάξουμε αν θέλετε αυτή την άποψη ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξει μια διεθνής συνθήκη για το αντίθετο, δηλαδή για την αποφυγή τέτοιου είδους πρακτικών. Εάν έρθει τελικά μια μέρα όπου θα δίνουμε οικονομικό κίνητρο για μεταμόσχευση οργάνων ή για δωρεά οργάνων, ε, θα ανοίξουμε πραγματικά το κουτί της Πανδώρας και θα κάνουν μεταμόσχευση οργάνων μόνο όσοι μπορούν να τις ε, πληρώσουν. Νομίζω ότι όταν υπάρχουν εκστρατείε ευαισθητοποίηση τη κοινή γνώμη, αυξάνεται ο αριθμό των δωρητών. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό και θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση σε εκστρατεία συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Εν πάση πτώση να κάνετε οτιδήποτε θέλετε εκτός από το να δώσετε οικονομικό κίνητρο ε, για τις δωρεές και τις μεταμοσχεύσεις. Παρόλο που διανύουμε τέτοιου είδους ε, ε, κρίση οικονομική αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι αυτό στο οποίο ήθελα να επιμείνω. Και δεύτερον, ως προς την κρίση και τις περικοπές. Είπατε στην πρώτη σας παρέμβαση ότι πρέπει να είμαστε δημιουργικοί, πρέπει να έχουμε φαντασία, πιστεύω κι εγώ. Όντως, πρέπει να είμαστε επινοητικοί και αποτελεσματικοί. Αυτό είναι ένα όμως και άλλο είναι το εξής. Με τις πολιτικές που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη που τελικά περικόπτουν ψαλιδίζουν το δικαίωμα στην υγεία με πρόσχημα την κρίση και προκειμένου να είναι αποτελεσματικά τα κράτη-μέλη θα περικόψουν προϋπολογισμούς παντού. Δηλαδή, δεν θα σας βοηθήσουν οι υπουργοί, εσάς κύριε Μαλά, όπου στη χώρα τους κάνουν τέτοιου είδους περικοπές. Από το Συμβούλιο πρέπει να βγουν μηνύματα προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή να περικοπεί το οτιδήποτε εκτός από το δικαίωμα στην υγεία. Εγώ αυτό πιστεύω. Και θα πρέπει να αξιολογήσουμε κάθε πρόγραμμα με βάση το βάρος που έχει στον προϋπολογισμό. Τι σημαίνει όμως αυτό. Θα πρέπει να διεκδικήσετε κύριε Υπουργέ περισσότερα, να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία για να πείτε στους υπόλοιπους υπουργούς ότι φτάνει πια. Δεν γίνεται να χρησιμοποιεί κανείς το πρόσχημα, την επίφαση της κρίσης για να καταστρατηγεί το δικαίωμα στην υγεία δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε τέτοιου είδου περικοπές στο δικαίωμα της υγείας αν μπορούσαμε πραγματικά ε, να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, την φοροαποφυγή ε, και όλα αυτά τα δεινά που μα ταλανίζουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, για το θέμα που παρουσίασες με τόσο πάθος. Ο Καρλ Χάινς Φλόρενς που ήταν στην αρχή του καταλόγου αλλά μπερδέψαμε τη σειρά. Ευχαριστώ. Ναι, ε, ακούω τον κύριο Υπουργό που τόνισε ε, την πτυχή που ανέφερε η Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ. Δεν θα ήθελα να σας μιλήσω για τα φάρμακα, διότι εγώ φοβάμαι τους ιατρούς και δεν είμαι ειδικό. Ε, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στην προληπτική ιατρική και ιδιαίτερα όσον αφορά το κάπνισμα. 18 ε, χρόνια ή περισσότερα ε, ε, έχω πίσω μου στο θέμα αυτό. Η πρόοδος όμως πηγαίνει αργά σε σαλιγκάρι άσχετα από το ποια προεδρία έχουμε ανα πάσα στιγμή. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω σχετικά με την προσέγγισή σας. Η Κομισιόν αναφέρεται σε νέο νομοθέτημα που έχει να κάνει με την επισήμανση ε, σημαντικό είναι να μην αρχίζουν να, το κάπνισμα οι νέοι. Ε, μπορεί να είναι δύσκολο να κόψουν το κάπνισμα οι πιο μεγάλοι, αλλά το να μην ξεκινήσει το κάπνισμα ε, οι νέοι είναι πολύ σημαντικό και θα μπορούσαμε να ε, αναπτύξουμε κάποια εργαλεία εδώ, για παράδειγμα όσον αφορά την επισήμανση. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς το θέμα της, των χημικών και η καπνοβιομηχανία μας, ε, μας κοροϊδεύει ουσιαστικά. Ε, ε, υπάρχουν σημαντικές βλάβες στην υγεία από τα χημικά που περνάνε από τον επινευστικό στον εγκέφαλο και επηρεάζουν το γενετικό υλικό. Και σημαντικό είναι λοιπόν να σταματήσουμε ε, την πρακτική αυτή και να έχουμε ρύθμιση σχετικά με τα χημικά. Δεν είναι εξίσου απολαυστικό ε, κάθε τσιγάρο, διότι ο καπνός είναι ε, φυσικό προϊόν. Ε, τι, πώς το βλέπετε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το ένα αφορά τη δωρεά οργάνων. Πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικό και σε επίπεδο Συμβουλίου να μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά την υπόθεση ότι μπορεί να δωρηθεί ένα όργανο. Ακόμα και αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει εκφράσει προηγουμένως αυτή την επιθυμία. Δεν μπορεί να εκφραστεί πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι θα ήταν διαθέσιμα περισσότερα από τα ένα όργανα όσον αφορά τη δωρά οργάνων. Διατηρώντα τη γενική αρχή που πιστεύω είναι αδιαφυσβήτητη, της δωρεά, δωρεάν παροχής του οργάνου. Το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω, στις κλινικές δοκιμές, όσον αφορά την αδειοδότηση για το εμπόριο φαρμάκων. Είναι μια φάση, όπως είπατε σωστά, αυτή που περνάμε, εξαιρετικά δύσκολη, χερίς. Υπάρχουν όμως και οι φαρμακοβιομηχανίες που ε, δεν κάνουν πολλά, θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα, πολύ μεγαλύτερη δραστηριότητα να έχουν όσον αφορά τα φάρμακα για σπάνιες ασθένειες. Ενώ αντίθετα, όπως υπενθυμίσατε εσείς, έχουμε μία μείωση των νέων φαρμάκων που διατίθεται στο εμπόριο. Εδώ υπάρχουν κάποιες προτάσεις και για τον ορίζοντα 2020. Προτάσεις για δραστική αλλαγή, για αύξηση της ποιότητας των κλινικών δοκιμών, αλλά με τεστ που δεν χρησιμοποιούν απαραίτητα ζώα. ό,τι μπορεί να γίνει, όπως μπορεί να γίνει και με τα βλαστοκύτταρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά και οι στατιστικές ε, είναι πιο ακριβείς. Και μπορούν να έχουν πιο στενή αναφορά στον άνθρωπο οι δοκιμές αυτές σε σχέση με τις δοκιμές που γίνονται στα ζώα. Χρειάζεται λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτό που λένε οι φαρμακοβιομηχανίες. Ο κίνδυνος που υπάρχει στην ανάπτυξη και να φτάσει κανείς στη φάση είναι αυτός που αποκλείει τη δυνατότητά τους να δεσμευτούν για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να αλλάξουν οι κλινικές δοκιμές αδειοδότησης και θα μπορούσε να είναι αύξηση της ασφάλειας αυτή αλλά και να μειώσει και το κόστος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Βικτόριο Πρόντι. Η Τάκμα Ροντ Πέρεντ με μια συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να επανέλθω στις ιατρικές αυτές συσκευές γιατί δεν μπορούσα να συμπεριλάβω όλα στο, στην πρώτη μου παρέμβαση. Εντάξει, το πιάσα αυτό που λέτε, δεν χαίρομαι με αυτό που λέτε, αλλά χαίρομαι τον τρόπο που το παρουσιάσατε. Ε, για την εισαγωγική σας δήλωση δεν ήμουν πολύ ενθουσιώδης, τα υπόλοιπα ήταν πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι θέλετε να κάνετε τη διαφορά. Ελπίζω να κάνετε τη διαφορά στις ιατρικές συσκευές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε σαφή διάκριση μεταξύ αδειοδότησης και κοινοποίηση πιστεύω ότι έχουν αξία και τα δύο. Και κάτι που δεν εξετάζεται ταυτόχρονα οι θετικέ συσκευέ. Μοναδική και πολλαπλή χρήσεω συσκευέ. Όταν είδα τον ορισμό μία χρήσεω, πολλαπλή χρήσεω, που πρέπει να υπάρχουν οι ορισμοί και μιλάμε για πολλαπλή χρήση, τότε μπορούμε να δούμε τα θέματα τη υγιεινή στα νοσοκομεία και στου διάφορου φορεί να υπάρχει μια συνεχής νομοθεσία για την υγεία, για την ανάκτηση και επανεπεξεργασία αυτών των ιατρικών συσκευών για πολλαπλή χρήση. Κατά την άποψή μου αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αποφύγουμε ε, τις μολύνσεις ε, στα νοσοκομεία και τα ιδιαίτερα ανθεκτικά βακτήρια που δεν έχουμε αρκετά αντιβιωτικά. Μήπως μπορεί να δοθεί και άλλο ένα κίνητρο για καινοτομία σε νέα αντιβιωτικά που καταπολεμούν ε, μολύνσεις που αντιστέκονται σε πολλά φάρμακα ε, που είναι κάτι που έχει πειράσει πολύ την, ε, το ιστορικό των ασθενών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο δεύτερος γύρος έκλεισε, οπότε έχετε τον λόγο να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Έχετε τον λόγο. So, I wasn't about the first question, Mr. Δεν είμαι σίγουρος για το πρώτο ερώτημα ε, του κυρίου Ροντρίγκες Έφυγε. Α, εδώ είσαστε. Σε αυτή την πρόταση δεν λέμε κάτι για οικονομικό κίνητρο. Ε, ίσως δεν, δεν με καταλάβατε. Αυτό που προσεγγίζουμε ε, δεν είναι αυτό στόχο. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε την κοινωνία και να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαίων. Αυτό είναι το πνεύμα της προσεγγίσεώς μας. Να αυξηθεί η κοινωνική ευαισθητοποίηση. Θυμηθείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Ακόμα και αν κάνετε σύγκριση σε παρόμοιε κοινωνίε. Πάμε την κοινωνία τη Κύπρου και την ελληνική κοινωνία. Συγκρίνετε την ανταπόκρισή του Η κοινωνική δέσμευση όσον αφορά τη δωρά οργάνων. Δείτε με τι γίνεται με το μυαλό των οστών. 200.000 δότες ε, και 50.000 στην Ελλάδα. Και ο πληθυσμό είναι 10 φορέ μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Άρα η κοινωνική κινητοποίηση και η κοινωνική ευαισθητοποίηση είναι το κλειδί θεμελιώδου σημασία. Βεβαίω υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ποιότητα και ούτω Και νομίζω ότι αν δούμε τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι βρίσκουμε. Και είναι άλλη μια συνιστόσα που θα πρέπει να εξεταστεί. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι διαδικασίες αξιολογήσεως ζωντανών δοτών διαφέρουν από χώρα σε χώρα και θα πρέπει αυτό να εξομαλυνθεί. Διότι αυτή είναι η προσέγγιση να εισαγάγουμε από, το, από την πλάγια πόρτα την ε, πώληση οργάνων. Το είδαμε αυτό όταν δεν γίνει σκληρή η νομοθεσία. Το λέω σαν Υπουργό Υγεία. Ανησύχησα κάποτε και στη δική μα εθνική νομοθεσία αυτό το φαινόμενο. Περικοπές στον τομέα της υγείας. Ίσως θα έπρεπε να έρθετε μαζί μας όταν θα επαγματευτούμε με το τρίο, με την Τρόικα όχι με, το τρίο, με την Τρόικα. Όπου πηγαίνουν αυτοί, ακολουθούν τεχνοκρατική προσέγγιση. Και η υγεία είναι ένα τομέα που καμιά φορά τον πειράζουν. Συμφωνώ μαζί σα, ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε περικοπέ στον τομέα τη υγεία σαν αυτό σκοπό, γιατί χρειάζεται να ισολογήσουμε τον προπολογισμό. Αυτό κάνουμε, βασικά. Ταυτόχρονα όμω πρέπει να πούμε ότι δεν μα εμποδίζει αυτό από το να είμαστε καινοτόμοι δεν μας σταματά από το να δούμε πώς δαπανούμε τα χρήματά μας στην υγεία και να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να ξοδέψουμε λιγότερα χρήματα. Σαφές παράδειγμα όπου η παρέμβαση μπορεί να γίνει και μιλώ σαν Υπουργό Υγείας εδώ. Στον τομέα των φαρμάκων λοιπόν, διάφοροι τρόποι, διαφορετικοί τρόποι χρήση από διάφορες χώρες επηρεάζουν πόσο πληρώνει κανείς για φαρμάκα. Είδα διαφορετικά συστήματα. Εμεί εφαρμόσαμε διαφορετικό σύστημα στη χώρα μου και μειώσαμε τις δαπάνες για τα φάρμακα σε σημαντικό βαθμό. Και δεν πειράζουμε καθόλου την καινοτομία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε. Δεν νομίζω ότι τώρα αυτή την εποχή θα πρέπει να κάνουμε σοβαρές περικοπές όπως είδα σε διάφορες χώρες. Κυρίως να κόβουν ένα μεγάλο κομμάτι από τον προπολογισμό για την υγεία γιατί θέλουν να ισολογήσουν τον προπολογισμό. Μπορεί να πει κανείς ότι κατά τη χρηματοστατική κρίση το βάρος στον τομέα της υγεία θα αυξηθεί και πιθανότατα θα πληρώσουμε το κόστος της πολιτικής μας στο εγγύ μέλλον. Α έρθουμε τώρα στον καπνό, κύριε Φλόρενς. Βέβαια δεν θα συζητήσουμε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, έτσι μου λένε τουλάχιστον, να εκφράσω όμως την άποψή μου. Χρειαστήκαμε 40 χρόνια νομίζω για να προσπαθήσουμε και, για, και να μαζέψουμε τις επιστημονικές αποδείξεις για να αποδείξουμε τώρα ότι αδιαμφισβήτητα ο καπνός και το κάπνισμα, το κάπνισμα μάλλον, το κάπνισμα ε, είναι βασικός παράγων που δημιουργεί το καρκίνο. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα όσον αφορά την οδηγία για τον καπνό που ελπίζουμε να επηρεάσει την κατάσταση. Θα επηρεάσει όμω μαζικά τη δημόσια υγεία και τον τομέα τη περίθαλψη. Εξαρτάται από το τι θα συμπεριλαμβάνει. Αν δούμε την όλη ιστορία, το ιστορικό, Γαλλία α πούμε. Οι Γάλλοι όταν εισήγαγαν πολύ ψηλή φορολόγηση, χωρίς να πειράξουν την ετικετοθεσία, μείωσαν δραματικά το επίπεδο, τα ποσοστά καρκίνου του πνεύμονος. Και το ίδιο ισχύει και στον Αμένο Βασίλειο. Ήταν ένα μέτρο αυτό λοιπόν που χρησιμοποιήθηκε. Τώρα αν θα έπρεπε να απαγορευτεί ή να μην απαγορευτεί ε, δεν θέλω να τοποθετηθώ. Ε, ζούμε στην πραγματική ζωή και αυτή είναι προσωπική άποψη. Ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να απαγορέψουμε τα πάντα και να τα βγάλουμε το σύστημα. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι σημαντικό. Όποια δράση και να ακολουθήσουμε, η τικετοθεσία, υψηλή φορολόγηση, θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Διότι είδαμε νέους που δυστυχώ αυτές τι μέρε έχουν λιγότερες φιλοδοξίες ε, στη ζωή τους ε, να εκτίθεται στο κάπνισμα περισσότερο. Από ό,τι κατάλαβα, η Ιρλανδική Προεδρία θα ασχοληθεί με το θέμα. Οι πρώτε αντιδράσει που είδα είδα κάποιο μήνυμα ότι ίσως να συζητήσουμε αυτή την οδηγία. Ακούγεται αυτό πολλού τομεί, πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν θα προκύψει. Κύριε Πρόντι, αναφερθήκατε στη δωρεά των οργάνων και τη σύμφωνη γνώμη, την έγκριση, συνένεση, ρωτάτε κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε πρώτερη συνένεση κάποιου ατόμου που είναι υποψήφιος να δωρήσει ένα όργανο, ένας ασθενής ο οποίος ε, προφανώς θεωρείται κλινικά νεκρός και δεν είχε δυνατότητα να εκφράσει τη συνένεσή του. Άρα θα πρέπει να αυξήσουμε τη δυνατότητα διάθεσης οργάνων αν ένα άτομο δεν μπορεί να δώσει τη συνένεσή του. Αυτό είναι θέμα κοινωνικό, γίνεται σε κάθε χώρα ε, και είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Κάποιες χώρες κατάφεραν πραγματικά να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα, να βρουν κάποια λύση. Ε, νομίζω ότι όσο πιο πολύ εμπλέξουμε την κοινωνία και όσοι πιο πολλοί δωρητές οργάνων υπάρχουν στις χώρες μας, τόσο θα, θα λύσουμε το πρόβλημα. Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Ποτέ δεν θα μπορέσει κανείς να το συζητήσει αυτό, διότι κάποιες κοινωνίες έχουν και θρησκευτική τοποθέτηση πολύ αυστηρή και δεν το επιτρέπουν όπως πιστεύω ότι το γνωρίζετε. Όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές, αμενεθήκατε και στην ε, καλλιέργεια των ε, κυτάρων. Ε, το θέμα των κυτάρων είναι θέμα επιστημονικό, κατά πόσο μπορούμε να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα όσον αφορά την αξιολόγηση των φαρμάκων σε ένα σύστημα καλλιέργειας κυτάρων σε αντίθεση με πλήρεις δοκιμές επί ή επιζών, ζώων, επί ανθρώπων ή επί Αν μιλήσω ως επιστήμον, νομίζω ότι πιθανότατα ποτέ δεν θα μπορέσει κανείς να αντικαταστήσει τις κλινικές δοκιμές με τα κύτταρα, με καλλιέργειες κυτάρων. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό και διατρέχει κάποιο τον κίνδυνο να δημιουργήσει ένα θεμελιώδε πρόβλημα. Πρόβλημα όσον αφορά την διάθεση στην αγορά των προϊόντων. Αυτό μπορεί να γίνει και γίνεται. Είναι αντί να χρησιμοποιήσουμε καλλιέργεια κιτάρων... να κάνουμε αυτό που είπα προηγουμένως, κοινέ πρωτοβουλίες τεχνολογικού περιεχομένου που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να κάνετε προσωμιώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, να χρησιμοποιήσετε κάποια καλλιέργεια κυτάρων και μπορείς να κάνεις δίθηση και να δεις ε, ποια φάρμακα μπορούν να είναι καλά για συγκεκριμένη ασθένεια. Έτσι μειώνεται το κόστος, διότι αναφερθήκατε και στη μείωση του κόστους, αλλά κατά την ταπεινή μου γνώμη ποτέ δεν μπορεί να αντικαταστήσει κανείς τις δοκιμές. Επανήθατε στο βασικό θέμα που σας αρέσει. Δεν είμαι σίγουρος τι εννοούσατε όσον αφορά το θέμα τα, τα εμφυτεύματα. Αναφερθήκατε σε καθόδες θέμα. Γιατί να μην σας στείλουμε γραπτός μια απάντηση, γιατί νομίζω ότι δεν έχετε πιστεί πολύ από την απάντησή μας, θα σας στείλουμε γραπτή απάντηση. Ο κύριος Πρόντι για μια σύντομη παρέμβαση, έχετε το λόγο. Βιτόριο δεν έλεγα να απαλλαγούμε από τις δοκιμές τα ζώα. Έλεγα όμως τα πειράματα όσον αφορά τις καλλιέργειες χιτάρων μπορούν να δώσουν λεπτομερέστερες απαντήσεις όσον αφορά τοξικολογικούς μηχανισμούς και μπορεί αυτό να ταιριάζει καλύτερα με τους ανθρώπους από ό,τι δοκιμές στους, ε, στα ζώα. Ε, νομίζω ότι αυτή την ανοιχτή προσέγγιση εννοούσα για την αλλαγή των κλινικών δοκιμών ούτως ώστε να έχουμε ακριβέστερες απαντήσεις και χωρίς να απαλλαγούμε βέβαια να μειώσουμε όμως τις δοκιμές στα ζώα. Απάντηση. Νομίζω Αναφερθήκατε σε προληπτική τοξικολογία. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζει η φαρμακοβιομηχανία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του IMI, για αυτούς που γνωρίζουν, την πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα, με άλλα λόγια, και πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία και πολλά χρήματα διατίθεται για την προβλεπτική, προβλεπτική τοξικολογία που δεν χρησιμοποιεί ζώα χρησιμοποιεί καλλιέργειες κιτάρων και προσωμιώτες σε υπολογιστές για να προβλέπονται οι τοξικολογικές συνέπειες των υποψηφίων ουσιών, των εξεταζομένων ουσιών. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τον ε, κύκλο ερωτήσεων και απαντήσεων και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, ιδιαίτερα θερμά τον Υπουργό Υγείας κύριο Σταύρο Μαλά για τις ε, αναλυτικές ε, και ε, πολύ καλές απαντήσεις του. Όπως είπαμε, είσαστε πολύ φιλόδοξος όσον αφορά την Προεδρία σας. Ε, μπορώ να το επιβεβαιώσω. Είχαμε συνάντηση στο γραφείο μου και εντυπωσιάστηκα πολύ από τις γνώσεις σας. Είσαστε ειδικό. Ο καθένας μπορεί να το διαπιστώσει αυτό αν διαβάσει το βιογραφικό του ε, Υπουργού. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ειδικό στα θέματα αυτά. Προσλέπω λοιπόν ε, στο επόμενο εξάμεινο στην Προεδρία της ε, Κύπρου. Μας κάνατε συγκεκριμένες προτάσεις και όπως είπε η συνάδελφος Ροτ Μπέρεντ, ε, να τονίσετε ιδιαίτερα την νομοθετική πτυχή. Είμαι πεπισμένος ότι ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης, ε, στις οποίες αμφισβήτητα βρισκόμαστε, μια καλή πολιτική υγείας ε, αποτελεί πολύ θετικό μήνυμα προς 500.000 Ευρωπαίους. ώστε να μπορεί ο καθένας από αυτούς να ε, να επωφεληθεί από την Ευρώπη και ε, να μην πληρώνει ε, το κάθε άτομο το τίμημα της κρίσης. Σας εύχομαι λοιπόν μια επιτυχημένη και φιλόδοξη Προεδρία. Είσαστε πάντα ευπρόσδεκτος. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Μετά λοιπόν από την παρουσίαση της ε, Προεδρίας του Συμβουλίου ξεκινάμε, ε, συνεχίζουμε την ε, εξέταση της μερικής διάταξης με το σημείο 5 λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης ε, για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων ε, που σχετίζονται με τις ε, χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομεία. Ο Κρήτον Αρσένης είναι εισηγητής, θα μας διαφωτίσει λοιπόν σχετικά με το θέμα αυτό. Κατόπιν θα προχωρήσουμε στην συζήτηση με τους κοιότητες. Παρακαλώ Κρήτον, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ να μην ε, ε, περιμένουν οι συνάδελφοι ότι θα τα εξηγήσω τόσο καλά όσο ο Υπουργός της ε, Κυπριακής Προεδρίας. Είναι μια πρόταση λοιπόν αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λογιστική καταχώρηση των χρήσεων γης, των αλλαγών χρήσεων γης και της δασοκομείας. Υπάρχει εδώ και κάποιους μήνες. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στο Μαρακές. Μάλιστα, δεν είναι μόνο κάποιοι μήνες, είναι πάρα πολλά χρόνια, γιατί το, στο το Μαρακές συνέβη, πριν, πριν, συνέβη το 2001. Όμως, πρόσφατα στο Ντέρμπαν υπήρξε τελική απόφαση για υποχρεωτική λογιστική καταχώρηση της διαχείρισης των δασών ούτως ώστε να είναι πολύ πιο ορατό το απόθεμα άνθρακα. Ποια είναι η πρόταση σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχουμε ομάδες για τη λογιστική καταχώρηση τέτοιων δραστηριοτήτων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναπτυχθούν αυτά τα σχέδια δράσης, ούτως ώστε να διαδοθούν οι πληροφορίες και τα στοιχεία στα κράτη-μέλη για τις εκπομπές που σχετίζονται με τέτοιου είδους δραστηριότητες. Η απόφαση αυτή είναι το πρώτο στάδιο της προσέγγισης δύο φάσεων. Δηλαδή, η βασική ιδέα είναι πια. Ξεκινούμε με την θέσπιση των κανόνων για τη λογιστική καταχώρηση, αυτή είναι η πρώτη φάση, και στη δεύτερη φάση υπολογίζουμε τις εκπομπές ε, σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει για την μείωση των εκπομπών. Συζητούμε λοιπόν τώρα τη φάση 1. Η απόφαση δεν επιβάλλει δεσμευτικούς στόχους, ούτε διατάξεις. Είναι ένα τεχνικό έγγραφο το οποίο θεσπίζει κανόνες για την ορθή λογιστική καταχώρηση παρόλο που όλα αυτά έχουν αποφασιστεί σε διεθνές επίπεδο. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο πόσο σοβαρά λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα οποία αποφασίζονται στις διαπραγματεύσεις ε, με τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές. Πόσο σοβαρά είναι αυτά τα οποία για τα οποία δεσμευόμαστε σε διεθνές επίπεδο. Και είναι και ένας πολιτικός συμβολισμός πολύ σημαντικός εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τη στιγμή που έχουμε το στόχο να ε, έχουν οι διαπραγματευτές μας μια συμφωνία που να έχουμε ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τη στιγμή που ε, στις αρχές του, Δεκεμβρίου ε, θα πάνε στην Τόχα για την ε, διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, το COP18 μπορούμε να πούμε ότι εκεί θα μπορούμε να πούμε ότι πριν από ένα χρόνο στο Ντέρμπαν αποφασίσαμε για το LULUCF για τη λογιστική καταχώρηση χρήσεων γης, αλλαγών χρήσεων γης και τασοκομείας και τώρα στην Τόχα το Δεκέμβριο έχουμε να σας ε, φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Στόχος λοιπόν είναι να τηρούμε τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, προσχωρήσει σε διεθνείς συμβάσεις. Αυτό είναι ένας πρώτος στόχος. Δεύτερο, θέλουμε να έχουμε συνεκτικότητα στην πολιτική μας, να έχουμε καλύτερο συντονισμό, ενοποίηση όλων αυτών των ε, στενοποίηση όλων αυτών το πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές οδηγίες. Και τρίτος στόχος είναι η πρακτική και μεθοδολογία να υπόκειται στις αρχές της διαφάνειας, της συνεκτικότητας, της συγκρισιμότητας, της ακρίβειας, όχι μόνο στο εσωτερικό των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των κρατών μελών. Τώρα, ως προς την υποχρέωση ε, καταχώρησης. Η υποχρέωση αυτή καταχώρησης σε σχέση με τις εκπομπές είναι πολύ σημαντικό βήμα, ούτως ώστε όλοι αυτοί οι τομείς να μπουν ε, στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. οποιοδήποτε είδος υποχρεωτική ε, λογιστική καταχώρηση θα είναι ουσιαστικά ε, άσκηση για τα κράτη-μέλη, για το πώς θα τηρούν τους κανόνες. Έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν την μεθοδολογία που εξηγείται στο κείμενο η οποία δεν διαφέρει από αυτή που ισχύει διεθνώ. Έχουμε αυτή την περίοδο 8 ετών τουλάχιστον για να υιοθετήσουμε αυτή τη λογιστική καταχώρηση μέχρι το 2020, επομένως έχουμε απλά το χρόνο να προετοιμαστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, έχει προτείνει ε, τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της λογιστικής καταχώρησης για τις εκπομπές σε σχέση με τους βοσκότοπους και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τη διαχείριση αυτών. Όλα τα κρατη έχουν ε, τα στοιχεία στη διάθεσή τους. Έχουμε τρία είδη στοιχείων το Peer 1, τα πιο απλά, τα πιο απλουστευμένα ως προς τη μεθοδολογία. Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνει μέχρι το Peer 3. Όλα τα κράτη-μέλη λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν από, την, από το πρώτο στάδιο και να προχωρήσουν σιγά σιγά προς το δεύτερο και το τρίτο. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά εξοπλισμένοι ως προς αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο πράγματι να εφαρμοστεί από όλους η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ προτείνω να συμπεριληφθεί και η αποστράγγιση και η επανήγρανση υγροτόπων ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της λογιστικής καταχώρησης εκπομπών είναι ο πιο κατάλληλος για το θέμα αυτό. Γιατί διότι στις ενδιάμεσες διαπραγματεύσεις για το κλίμα και τις κλιματικές μεταβολές και τη συνθήκη αυτή, εδώ στο Κοινοβούλιο το είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό. Ε, υπήρχε ένα θέμα οργάνωσης, αν θέλετε. Ήταν όλοι σε μια άλλη αίθουσα στην αρχή, όπου εκτιλήσονταν οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τους νέους λουλογιστικούς κανόνες για την καταχώρηση αυτή. Συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση των κανόνων και όπως ξέρετε αυτοί οι κανόνες για τη λογιστική καταχώρηση τώρα τίθεται ε, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιώτο, όμως μέχρι το 2015 ε, θα επιτευχθεί νέα συμφωνία η οποία θα ισχύσει μέχρι και το 2020 στην οποία θα υποχθεί αυτή, αυτή η λογιστική καταχώρηση. Σε αυτή τη συμφωνία θα, θα προσχωρήσουν και οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλες χώρες και ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουν συμπεριληφθεί ε, και οι υγρότοποι και η αποστράγγιση αυτών και η επανήγρηση, η γράνση αυτών. Επομένως θα είναι ένα νέος τομέας, ένα νέο πεδίο συνεργασίας. Όπως και στο παρελθόν, ό,τι είχε να κάνει με τη δασοκομεία δεν είχε, δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα. Το ίδιο ε, θα συμβεί και εδώ πριν το 2020 θα καταστεί υποχρεωτικός ο χαρακτήρας αυτός για τους ε, υγρότοπους πριν να ε, λήξει η περίοδος ισχύως από, για αυτές τις αποφάσεις. Υπάρχει μία εξαίρεση για εκπομπές από δάσωση και δραστηριότητε διαχείρισης των δασών σε κάποιες περιστάσεις. Ποια είναι η ιδέα. Αν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα ή κάποια φυσική καταστροφή, τεράστια πυρκαγιά που καταστρέφει πάνω από 5% του δάσους μιας χώρας, που συμβαίνει ισπανιότατα βέβαια, τότε οι εκπομπές που προέρχονται από αυτή την πυρκαγιά μπορούν να εξαιρεθούν. Η προσήγγιση μου στο προτινόμενο σχέδιο εκθέσεως που έχετε μπροστά σας είναι να επιστρέψουμε στο κείμενο που αποφασίσαμε στο Ντέρμπαν για να υπάρχει συνέπεια. Αν έχετε ερωτήσεις, με τα χαράς να συζητήσω μαζί σας. Τώρα τα προϊόντα ξυλίας από υλοτομία. Τι είχαμε αποφασίσει. Όταν κάνουμε υλοτομικέ δραστηριότητε και χρησιμοποιούμε την ξυλία για έπιπλα, ή άλλα προϊόντα ξύλινα. Θεωρούμε τα έπιπλα να είναι κάτι πράγμα, κάτι νεκρό. Ε, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει άλλη οξύδωση περαιτέρω και εκπομπή κάποιο για τα ξύλινα προϊόντα, για τα έπιπλα. Υπάρχει κάποια χρονική καθυστέρηση όσον αφορά την εκπομπή του άνθρακος. Και αυτό προστίθεται στην νομοθεσία. Το θέμα είναι τι συγκεκριμένα στοιχεία χρησιμοποιούμε για να αντικατοπτήσουμε αυτά, αυτά τη μισή διάρκεια ζωής όσον αφορά τον άνθρακα στα έπιπλα και άλλα ξύλινα προϊόντα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα ειδικά στοιχεία άλλου κράτους και για εισαγωγέ. Φανταστείτε λοιπόν. Η Γερμανία και η Γαλλία εισάγουν ξυλία από τη Ρωσία ή από το Βέλγιο. Χρησιμοποιούν την εκτιμόμενη μίσια ζωή, την τιμή μίσια ζωής για την ξυλία που εισάγουν και έπιπλα και ξύλινα προϊόντα που εισάγουν από το Βέλγιο με διαφορετικό τρόπο. Η γερμανική εκτίμηση διαφορετική από τη γαλλική. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για τη συνέπεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, για αυτά τα προϊόντα από ξυλία, από πελοτομία, απαιτείται κάτι μέλλον και να μπουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αναθεώρηση να χρησιμοποιήσουν κατά χώρα η μίσια διάρκεια ζωής για την εξαγωγή ξύλινων προϊόντων, προϊόντων ξυλίας εκτός της Ένωσης και να απαγορεύει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ειδικέ διάρκειε ημίσια ζωή για τα είδη ξυλία που ετίθονται εντό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που παρεκκλίνουν από αυτά που χρησιμοποιούν τα εισάγοντα κράτη-μέλη. Επίσης, ένα θέμα βασικό για τις συζητήσεις μας. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Διότι κατά κράτη μέλη και, ε, και οι συνάδελφοι εξέφρασαν αμφιβολίες όσον αφορά τα διάφορα σχέδια δράσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια λογική πρόταση. Κάποιοι θεώρησαν ότι υπήρχε πρόβλημα με την επικουρικότητα και ότι υποχρεώνονται να εφαρμόσουν κάποιε πολιτικέ τα κράτη-μέλη. Εξαρτάται πώ ερμηνεύει κανεί τα γραφόμενα και όχι τα γραπτά αυτά κάθε αυτά. Γι' αυτό η ερμηνεία οδηγεί στο να ανησυχούν κάποιοι και νομίζω ότι είναι απλούστατα τα πράγματα. Έκανα κάποιες προτάσεις διατύπωσης αναφερόμαστε στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών. Και πρόσθεσα και κάποια κείμενα, κάποιες διατυπώσεις για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Τα σχέδια δράσης ε, είναι η ανταλλαγή ε, πληροφοριών όσον αφορά τις εκπομπές από δεσιότητες των κρατών μελών και τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για τη μείωση των εκπομπών. Χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών, διότι δεν έχουμε άλλη πηγή ε, τέτοιων πληροφοριών την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η συμμετοχή του κοινού αναφέρεται εδώ, η διαφάνεια, κάτι που απαιτείται και σε άλλα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χρειάζεται και εδώ. Κλείνοντας, αναφέρομαι στους ορισμούς. Αρκετοί όροι που χρειάζονται στο έγγραφο χρειάζονται διευκρίνηση, ε, δεν έχουν οριστεί. για αποθήκευση, αποδάσωση, αποψήλωση, τα προϊόντα ξυλίας κλπ. Διάφορους όρους τους διευκρινίζω καλύτερα. Όπως ε, στιγμία οξύδωση κλπ. Για τον ορισμό των δασών, πολλοί συνάδελφοι το έθεσαν. αμφισβητήσιμο θέμα εδώ. Ποιο είναι το πρόβλημα. Εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουμε στην ΚΑΠ ορισμό για τα δάση. Είναι πιο στενός από τον παγκόσμιο ορισμό. Περιγράφει πιο στενά το τι είναι δάσος από ότι από το UNFCCC. και βρήκαμε εδώ τρόπο να μειώσουμε τις εκπομπές μας σε αυτόν τον ορισμό. Και οι πόροι προέρχονται την κοινή αγροτική πολιτική. Αν βάλουμε στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στοιχεία του ευρύτερου ορισμού που αποφασίστη ε, από τα κάτω μετέχουν τις αποφάσεις ε, του COP στην Τέρμπαν στο Ντέρμπαν. Αν το κάνουμε αυτό θα έχουμε κανόνες λογιστικού υπολογισμού για να μετρήσουμε και να μειώσουμε τον, τις εκπομπές βασιζόμενοι σε ευρύτερο ορισμό από αυτόν που χρησιμοποιούμε ε, στο εσωτερικό για να χρηματοδοτούμε τη μείωση των εκπομπών. Αν έχουμε τον ορισμό του ΚΟΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην απόφαση LUCF τότε υπάρχει συνέπεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εφόσον χρησιμοποιεί ορισμό που είναι στενότερος από τον άλλον, την απόφαση LUCF-COP, συμμορφωνόμεθα και με τα όσα κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Σωστή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ευθυγραμμιστεί ο ορισμός αυτός με τον COP της γεωργικής ε, πολιτικής η νομική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε αυτή την πρόταση, τη βρίσκω λογική. Εδώ θα σταματήσω και βεβαίω θα δώσω απαντήσει σε τυχόν ερωτήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κρήτονα. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδει εισηγητές. Η κυρία Μοκονάιτε είναι πρώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το έγγραφο Λουλουσιέφ είναι πολύ σημαντικό υπό το φως της παρούσας πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλλαγή του κλίματος και νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε κοινή θέση πάνω στο θέμα αυτό. Είμαι ευγνώμων στον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει καθώς και απέναντι στην Επιτροπή που υπέβαλε την αρχική πρόταση που μας επιτρέπει να διεξάγουμε τη συζήτηση εδώ. Θα ήθελα όμως να θίξω κάποιες ε, ανησυχίες της πολιτικής μου ομάδας. Καταρχήν ε, το έγγραφο αυτό ακολουθεί τις γραμμές ε, που υιοθετήθηκαν πέρσι στον Τέρμπαν. Ε, κανείς ε, δεν αμφισβητεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να εκπονήσει κοινή πολιτική. Οι συζητήσεις που βλέπουμε κάθε χρόνο αφορούν τα ίδια θέματα. Η Κομισιόν πολύ σωστά υποβάλλει φιλόδοξες προτάσεις Χωρίς αυτό θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο να πετύχουμε κάποιους στόχους. Ε, έτσι έχουμε ένα ενέργεια για τις συζητήσεις, αλλά, είναι πολύ, αλλά πολύ σωστά ο εισηγητής προτάνει ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την πραγματικότητα. Ε, τα, ε, τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά συμφέροντα, ε, έχουν ακόμα και διαφορετικά δάση. Δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει τα δάση της Βόρειας Ευρώπης με της Νοτιού Ευρώπης. Ταυτόχρονα δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει τα δάση της Βορείου Ευρώπης καθώς και τα λογιστικά συστήματα για τις ε, γεωργικές χρήσεις με αυτά της Ανατολικής ε, Ευρώπης, ε, όπου υπάρχει σύστημα μόλις από το 1998. Δεν θα πετύχουμε, πιστεύω, θετικό αποτέλεσμα εάν οθήσουμε τα κράτη-μέλη να, να δεσμευτούν ακόμα περισσότερο ή προσπαθώντας να είναι πιο φιλόδοξα από ό,τι μπορούν. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε περισσότερες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πιο φιλόδοξο ε, κείμενο, παρότι υπάρχουν διαφορετικές ε, θέσεις για το θέμα αυτό. Επίσης, ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη επαρκώς η αρχή της επικουρικότητας και να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη όσον αφορά την υλοποίηση της συμφωνίας αυτής. Και επιτρέψτε μου να θέσω κάποιες ερωτήσεις, να ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον εισηγητή για συγκεκριμένα θέματα. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον ορισμό του δάσους, ο Κρήτον ήδη ανέφερε τον ορισμό της ανάπτυξης της υπαίθρου. Και ζητήθηκε αυτό το μισό εκτάριο ε, με βάση αυτό. Ωστόσο, ε, τα δάση ορίζονται διαφορετικά σε, ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Κάποιοι εφαρμόζουν 0,1 εκτάριο, άλλοι άλλα νούμερα. Τίθεται λοιπόν το θέμα πώς... Πόσες ε, αλλαγέ θα πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Το άλλο θέμα είναι όσον αφορά την επιλογή των συστημάτων ε, λογιστικής. Η Κομισιόν λέει ότι είναι αρκετά ευέλικτο το σύστημα, ωστόσο θα μπορούσε ενδεχομένω να μα δώσει περισσότερε εξηγήσει, διότι νομίζω ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν ανησυχίε σχετικά με το σημείο αυτό. Άλλο θέμα είναι η συνέπεια όσον αφορά τις ε, απαιτήσει ε, στο πλαίσιο της LULUCF ε, και στα πλαίσια άλλων οργάνων του ΟΗΕ. Μήπως υπάρχει επικάλυψη και θα έχουμε υπερβολική γραφειοκρατία όσον αφορά το σύστημα υποβολής εκθέσεων. Και άλλο ενδιαφέρον θέμα για την δική μας ομάδα είναι η συμπερίληψη της γεωργικής γης. Ε, πιστεύω ότι αυτό καταρχήν ε, αντικρούει στο θεματολόγιο της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, και επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις επιθυμίες των κρατών μελών. Πιστεύω ότι θα ήταν δυνατότητα να διαχωρίσουμε τις γεωργικές εκτάσεις από τους βοσκότοπους. Από ό,τι κατάλαβα στον Τέρμπαν, η διατύπωση ήταν ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να υιοθετήσουν την πρόταση αυτή. Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, ε, σημαίνει ότι πρόκειται για προαιρετικό λίγο πολύ μέτρο. Και, ε, και μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Πιστεύετε και δέχεστε ότι τα ε, προαιρετικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον είναι προαιρετικά στο πλαίσιο του ΕΟΓΕ, δηλαδή να μην προχωρήσουμε περαιτέρω εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να διατηρήσουμε τις ε, υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που ήδη έχουμε σε διεθνές επίπεδα, απέναντι σε διεθνείς οργανισμούς. Και ε, να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο καινούριο στο σύστημα αυτό. Τα κράτη-μέλη ήδη υποβάλλουν τις σχετικές εκθέσεις. Ε, και μπορεί να έχουν διαφορετικά είδη δεδομένων, αλλά υπάρχουν κάποια ερωτήματα για τους ε, γεωργούς, για τον σχετικό κλάδο στα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχουν ερωτήματα λοιπόν σχετικά με το τι σημαίνουν όλα αυτά. Μήπως ε, μπορείτε να μας το διευκρινίσετε αυτό. Εμείς ερμηνεύουμε την πρόταση όταν τη διαβάζουμε. Εάν λοιπόν υπάρχει περιθώριο ερμηνείας ίσως να μην είναι απόλυτα σαφές ε, τι σημαίνουν όλα αυτά στην πραγματικότητα. Αυτά, αυτές κατά βάση είναι οι ανησυχίες μου και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο για να το συζητήσουμε. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ε, τις ανησυχίες μου αυτές. Περιμένω λοιπόν να λάβω απαντήσεις και διευκρινήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος με για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο αλλά και τον Κρήτονα γιατί έχει κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Νομίζω ότι κάποια από τα πράγματα που ακούσαμε είναι καταπληκτικά. Το LULUCF πράγματι θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος και θα βοηθήσει ώστε να αποφευχθούν ή να μετριαστούν οι κλιματικές μεταβολές. Είναι πολύ σημαντικό ως Κοινοβούλιο να ε, το δηλώσουμε αυτό και να ε, το προσυπρογράψουμε. Σε κάθε περίπτωση υψώνονται μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας, αν πραγματικά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές μεταβολές. Όντως, πάρα πολλά στοιχεία λείπουν ε, από την έκθεση. Δεν ξέρω αν γίνεται δίκαιη η αντιμετώπιση ε, της δασοκομείας παντού στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει αρκετή έρευνα, ούτε νομίζω ότι έχουμε εμβαθύνει αρκετά πάνω σε αυτό, μέσα σε αυτό το ζήτημα. Είναι σημαντικό. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο Ντέρμπαν να μπορούν να εφαρμοστούν σωστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μακροπρόθεσμα μάλιστα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκλίνει αρκετά από τη διεθνή συμφωνία που έχει επιτευχθεί για το θέμα αυτό. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω ότι ε, βρίσκουμε πολλούς λόγους ανησυχίας. Καταρχάς τα σχέδια δράσης δεν θα ήθελα να επικρίνω αυτές τις προτάσεις για τα σχέδια δράσης. Κατά την άποψή μου, το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι οι διαφορές είναι μεγάλες στην εκάστοτε πολιτική διασωκομεία και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η διασωκομεία στο βορρά και που ενδεχομένως μπορεί να γίνεται στο νότο. Για αυτό το λόγο λοιπόν είναι μεγάλο βήμα τελικά να έχουμε ένα σχέδιο δράσης που να εφαρμόζεται παντού στην Ευρώπη σε όλους τους εθνικούς κλάδους εθνικής δασοκομείας. Δεν νομίζω ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίζει από μόνη της για τη δασοκομεία και για το πώς θα χρησιμοποιούμε εμείς τα δάση μας και πώς θα τα αξιοποιούμε. Τώρα, όπως και η προηγούμενη ομιλήτρια, πιστεύω ότι οφείλουμε να εμείνουμε στη γραμμή που αποφασίστηκε στον Τέρμπαν. Αυτή είναι η δεύτερη μου παρατήρηση. Και η τρίτη μου παρατήρηση έχει να κάνει με τα στοιχεία που παρατίθενται εδώ. Έχουμε τα σημεία αναφοράς, τους αριθμούς που λειτουργούν ως σημεία αναφοράς. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα που κάνουμε προς μία ενιαία πολιτική για τη δασοκομεία. Και θα έλεγα επίσης ότι μπορεί κανείς να αντιληφθεί πλήρως την κατάσταση αν εξετάσει τα εθνικά αριθμητικά στοιχεία και τον τρόπο με τον οποίο έχουν μεταβληθεί. Νομίζω ότι ε, στην έκθεση αυτή και στις τροπολογίες ενδεχομένως ε, πηγαίνει το πράγμα πιο πέρα από ό,τι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είμαι βεβαία κατά πόσο μπορούμε να υποστηρίξουμε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής αυτής της έκθεσης ώστε να καλύψει και άλλους τομείς επίσης. Νομίζω ότι έχουν γίνει μεγάλες προσαρμογές στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον εισηγητή, ωστόσο χρειάζονται ε, να συζητηθούν κάποια θέματα ακόμα περισσότερο. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος ε, Τζούντι Κέρλινγκ μας είπε ότι επειδή έχει μια δέσμευση, μήπως μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά. Τη είπα μόνο εάν συμφωνούν οι συνάδελφοι. Βλέπω ότι ε, συμφωνεί ο συνάδελφος. Παρακαλώ, Τζούλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομη. Ήθελα να πω ότι ευχαριστώ τον εισηγητή για τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει. Ίσως όμως ε, έχει υπερβολική φιλοδοξία. Και εγώ θα ήθελα να σχολιάσω σε πιο πρακτικό βαθμό τα θέματα. Πράγματι πρέπει να ευθυγραμμίσουμε το κείμενο με τον Τέρμπαν και θα υποβάλω τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν συμφωνώ όμως να προχωρήσουμε περισσότερο από ότι τον Τέρμπαν. Αυτό θα προκαλούσε σύγχυση κατά την άποψή μου. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς συμφωνίες αλλά να μην τις ξεπερνάει γιατί ιδελώς υπονομεύουμε την δυνατότητα εφαρμογής της πρότασης. Ως προς τις πράξεις κατεξουσιοδότηση, ως προς το άρθρο 4 και 6 νομίζω ότι είναι κάτι το υπερβολικό. Ε, ενδεχομένως να έχει οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις οποιαδήποτε αλλαγή στα άρθρα αυτά, άρα να γίνει η αλλαγή αυτή για τις συνήθους διαδικασίες και όχι για τις διαδικασίες της επιτροπολογίας. Αυτή είναι η απόψή μου. Τώρα, ως προς τα εθνικά σχέδια δράσης, πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να μειωθεί το βάρος για ορισμένα κράτη-μέλη, να, είναι πιο ε, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη χρονική προθεσμία και θα υποβάλω τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ως προς τη διαχείριση βοσκότοπων και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, συμφωνώ με τους Ραντ Βίλερ Ίσως είναι υπερβολικό η Επιτροπή να θέλει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των καταχωρήσεων ε, για τις, ε, τους βοσκότοπους και την ε, καλλιεργήσιμη έκταση. Εγώ θέλω να επανέλθει ο εθελοντικός χαρακτήρας. Επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κρίμα, Τζούλη, που θα χάσετε τη δική μου παρέμβαση αφού πρέπει να φύγετε, αλλά τι να γίνει. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του. Οφείλω να πω ότι σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε με τις προτάσεις σας, ωστόσο, σε αντίθεση με την Τζούλη, η οποία φεύγει μόλις τώρα από την αίθουσα, εγώ δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξος ο εισηγητής. Μάλιστα πιστεύω ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξος. Με εκπλήσει το γεγονός ότι όλοι στο Κοινοβούλιο θέλουν να ευθυγραμμιστούν με τη Συμφωνία Ντέρμπαν, ενώ ξέρουν ότι θα αλλάξει σίγουρα του χρόνου και αν όχι του χρόνου, σίγουρα το 2015. Επομένως, μόλις υιοθετήσουμε τελικά αυτό το σύστημα, τότε θα ξαναξεκινήσουν και θα προχωρήσουν οι διεθνείς διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να ξαναλλάξουμε την νομοθεσία μας. Θυμάμαι ότι πάντοτε το Κοινοβούλιο ήθελε να είναι μπροστά, όχι να κυνηγάει από πίσω αλλά φαίνεται ότι τώρα το πνεύμα που διέπει το Κοινοβούλιο είναι ας ακολουθήσουμε τους υπόλοιπους, ας μείνουμε τελευταίοι στην ουρά. Ε, εγώ, εμένα αυτό με λυπεί και δεν νομίζω ότι θα πρέπει αυτό το πνεύμα να μας διέπει. Εν πάση περιπτώσει, στον οδικό ε, χάρτη ε, για το τον οδικό χάρτη για τις χαμηλές κουμπομπές δικαιοξυδίου του άνθρακα, στον, για τον οποίο συμφωνούμε όλοι, εκτός από το Συμβούλιο, υπογραμμίζεται ότι η χρήση γης είναι θεμελιώδες για την επίτευξη του στόχου αυτού. για την επίτευξη όλων αυτών των μακροπρόθεσμων στόχων σε σχέση με τις χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση των χρήσεων γης η οποία θα παρουσιαστεί με την πρόταση αυτή. Μα είναι μια πρόταση για τη λογιστική καταχώρηση. Δεν είναι μια συνολική πρόταση για το τι θα κάνουμε επιτέλους με τις χρήσεις γης. Παρόλο που είναι μόνο πρόταση για τη λογιστική καταχώρηση, υπάρχουν συνάδελφοι που πιστεύουν ότι είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι. Τι να γίνει, λυπούμε γι' αυτό. Εγώ συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή. Πιστεύω ότι όλα αυτά είναι εφικτά. Και μάλιστα και με τη Φιλανδία. Τώρα, να σχολιάσω τα εθνικά σχέδια δράσης τα οποία έχουν εθελοντικό χαρακτήρα και προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβάλλει στην κατάρτιση εθνικού σχεδίου δράσης, το οποίο είναι ένας πολύ ήπιος τρόπος, εν προσέγγισης του θέματος. Νομίζω ότι πρέπει να τα συνδέσουμε τα εθνικά σχέδια δράσης με ε, τον οδικό χάρτη για τις χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και νομίζω ότι πρέπει εμείς να θέσουμε ήδη σημεία αναφοράς, επίπεδα αναφοράς και να πούμε ότι δεν θα πρέπει η κατανομή της χρήσης γης να αλλάξει, γιατί αν τελικά ε, πάμε σε ακόμα πιο χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τη χρήση γης, ε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το θέμα. Επαναλαμβάνω ότι μιλούμε μόνο για λογιστική καταχώρηση και για τους υγρότοπους. Έχει έρθει πλέον η ώρα να αρχίσουμε να, να καταχωρίζουμε. Τώρα, ως προς τα υλοτομημένα προϊόντα ε, ξυλίας, ασκείται πίεση για λόγους ε, ε πηγών ενέργειας βιοκαυσίμων και ούτω καθεξής. Και πρέπει να σκεφτούμε όλες αυτές τις ειδικές τιμές χρόνου υποδιπλασιασμού. Για όλα αυτά, σε όλα αυτά συμφωνώ με τον εισηγητή. Ως προς την εθνική όχληση, τις εθνικές όχλησεις πράγματι πρέπει να γίνεται reporting, να αναφέρεται όταν ξεπερνούν οι εθνικές όχλησεις το 5% τουλάχιστον σε Γενικέ γραμμέ, λοιπόν εκφράζω τη στήριξή μου στον εισηγητή και α προσπαθήσουμε να γίνουμε κάπως πιο φιλόδοξοι έτσι ώστε στο διεθνέ στερέωμα να πάρουμε για άλλη μια φορά τα ενία, να ηγηθούμε ξανά γιατί το Τέρμπαν δεν θα κρατήσει πολύ. Υπάρχει ζωή και μετά τον Τέρμπαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μπάσο, Κάλχαρτς Φλόρενς, μετά το Λίζε. Ε, είναι πάντα δύσκολο όταν οι ε, συνάδελφοι διαφωνούν, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να παραμένουμε ευγενικοί. Ε, πάντως έχω πιο ε, χαλαρή εντύπωση αφού του μίλησα με την ε, Κομισιόν. εγώ πιστεύω ότι το Λούλου είναι μηχανή του διαβόλου και θα σας πω γιατί η Κομισιόν κρύβεται πίσω από το ότι ε, θα πρέπει πρώτα να συλλέξουμε δεδομένα και να δούμε μετά πώς θα προχωρήσουμε. Ένας από τα ανάτοτα στελέχη της Κομισιόν ε, είναι ειδικό και θα ήθελα πολύ να ε, μου περιγράψει τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα δάση που υπάρχουν. Και το είπε αυτό η συνάδελφος ε, και από το ΕΛ. Και θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι ε, κάνουν με τα δεδομένα αυτά, πώ τα αξιολογούν και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα των δεδομένων αυτών που συλλέγουμε. Το άλλο που δεν καταλαβαίνω από την Κομισιόν στον τομέα του περιβάλλοντος είναι γιατί δεν έχουν τα δεδομένα. Εγώ είμαι αγρότης. Και κάθε χρόνο Μέχρι και για κάθε ε, τετραγωνικό μέτρο θα πρέπει να υποβάλω δεδομένα ε, τι κάνω στην εκμετάλλευσή μου, ε, γιατί και πώς. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σωστό. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει 33 δισεκατομμύρια θα πρέπει να γνωρίζει τι γίνεται με όλα αυτά. Ξέρει λοιπόν πολύ καλά πόσα εκτάρια έχω και πόσο ε, παλαιά είναι τα δέντρα η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας γιατί δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα δεδομένα αυτά ώστε να μην χρειάζεται να καθόμαστε εδώ πέρα να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Κάποιοι υπερβάλλουν θα μου πείτε όπως στη δικιά μου χώρα ενώ άλλες χώρες δεν έχουν καν κτηματολόγιο Εξήγησέ μου λοιπόν, σε παρακαλώ. Σε συμπαθώ πολύ. Μου, ε, είσαι πολύ συμπαθή συνάδελφο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πει πώ θα καταλήξει σε συγκεκριμένα νούμερα και κατόπιν να δούμε πώ θα προχωρήσουμε. Ε, και μια ερώτηση προ την ε, Κομισιόν. Έχουμε την ε, διασταυρούμενη συμμόρφωση, cross-compliance. Ε, ε, μαζί με την Dagmar καταφέραμε να περάσουμε τον κανονισμό για τα λοιπάσματα, τον κανονισμό για, τα, για την προστασία των φυτών. Κάποιοι πιστεύουν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηροί, αλλά παρόλα αυτά τον έχουμε. Έχουμε τη χλωρίδα, την πανίδα και τους βιότοπους. Θα πρέπει να εξηγήσω πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε μια χώρα, όσον αφορά την ε, υλοποίηση, ανάμεσα στην Ιταλία, μια χώρα που αγαπώ πολύ, και την Γερμανία. Χρειάζεται να σε εξηγήσω τις διαφορές. Έχουμε κανόνες ε, δασοκομείας. Δεν καταφέρνουμε ούτε να σβήσουμε τις ε, μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη και θέλουμε να ρυθμίσουμε κάθε τετραγωνικό μέτρο στην Ευρώπη. Εγώ φοβάμαι αν και οι δύο συνάδελφοι που πήραν τον λόγο πριν από μένα, ο ένας από αυτούς ήδη έχει φύγει, ε, ε, σαν άνθρωποι με πείθουν, αλλά όσον αφορά το, την ουσία δεν με πείθουν. Η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει επιτέλους να πάρει θέση. Ε, θέλει να υποστηρίξει αυτά που θέλουν ο εισηγητής και ο πράσινος ε, συνάδελφος. Ε, εγώ στην Κομισιόν ε, θα έλεγα κάτι άλλο. Θέλει να επανισάγει τη γραφειοκρατία και εγώ ως Γερμανός δεν έχω καμία κατανόηση για τη θέση αυτή. Και γι' αυτό θα δείτε εδώ την πικρή μου αντίσταση, αλλά λέω ρητά ότι ε, η γεωργία θα πρέπει να συμβάλλει ε, όσον αφορά το θέμα του διοξιδίου του άνθρακα. Δεν θα το κάνει αυτό ε, από μόνη τη, γι' αυτό θα πρέπει και εμείς να σπρώξουμε. Ευχαριστώ πολύ, Καλχάρη Φλόρενς. 11 Οκτωβρίου θα ασχοληθούμε με το θέμα της μείωσης της γραφειοκρατίας. Έχω καλέσει τον δόκτωρα Έντμουν Στόιμπερ στην Επιτροπή μας θα μπορέσει να μας αναφέρει πολλά παραδείγματα ε, το τομέων όπου έχουμε ε, δημιουργήσει τεράστια γραφειοκρατία όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, μεταφορά, την εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Οριζοντίως λοιπόν δεν υπάρχει καμία ανταλλαγή απόψεων αλλά φαίνεται ότι ε, ούτε στην Κομισιόν ε, υπάρχει. Ε, τη στιγμή που ο αγρότης Φλόρενς πρέπει να υποβάλει ένα σωρό στοιχεία και η Γενική Διεύθυνση του Περιβάλλοντος δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. 11 Οκτωβρίου λοιπόν θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. με το θέμα της εφαρμογή και ξέρω ότι Κάλχανς είναι ένα θέμα που αγαπά ιδιαίτερα. Ε, θα ασχοληθούμε λοιπόν πιο εντατικά με το θέμα αυτό. Επόμενος ομιλητή ο Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Κρήτονα για την έκθεση αυτή και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Ραντβίλε ε, ε, Μοκονάτη για την παρουσίαση της θέσης ε, του ΕΛΚ. Φυσικά θα ήταν επιθυμητό η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τόχα να υποβάλει απόφαση, αλλά είναι πολύ φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα και ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι ήδη με το πακέτο ε, κλίματος ε, και ενέργειας ε, με το ζόρι υπερψήφισαν και Νομίζω ότι με όλο το σεβασμό ε, δεν είναι τόσο σημαντικό το θέμα αυτό που έχουμε μπροστά μας. Ε, οι εξελίξεις στην Τόχα δεν θα, ασχοληθούν, ε, δεν θα εξαρτηθούν από το πόσο έχουμε προχωρήσει στο θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που απαιτείται. Άλλωστε νομίζω ότι υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις. Οι γεωργοί φοβούνται περισσότερη γραφειοκρατία, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε αναλυτικά το θέμα προτού να γνωρίζουμε τι συνέπειες θα έχει το θέμα. εγώ δηλαδή, δεν δηλαδή, διστάζω να το περάσουμε γρήγορα το θέμα αυτό. Νομίζω ότι περισσότερος χρόνο θα ήταν χρήσιμος. Γενικά πρέπει να ε, αναγνωρίζουμε ότι το θέμα του LULUCF ε, ε, θα ελαφρύνει κάπως το κόστος του κλίματος. Με την LULUCF το κόστος αυτό θα μειωθεί κάπως και γι' αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία, θα πρέπει όμως ε, αναλυτικά να εξετάσουμε το θέμα και να αποφύγουμε την επικάλυψη εργασιών και την ε, γραφειοκρατία. Θα ήθελα η Κομισιόν να μου επιβεβαιώσει ότι ε, η πρόταση αυτή δεν θα επιβαρύνει τον κάθε ατομικό αγρότη. Όπως ο Καλχάνς Φλόρενς, όλοι οι αγρότες πρέπει να υποβάλουν στοιχεία σχετικά με την χρήση γης. Ε, εάν ε, λοιπόν ισχύει αυτό, η Ρατβίλε Μοκουνάιτε είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, εργασία μετάφρασης μετατροπής. Αλλά δεν θέλουμε επιπλέον γραφειοκρατικό άχθος για τους αγρότες ή για τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να γίνει επεξεργασία των στοιχείων που ήδη συλλέγονται και να υποβληθούν στην Επιτροπή. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε τι κάνουμε με τα δεδομένα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους γεωργούς, ε, κίνητρα να κάνουν θετικά πράγματα για το κλίμα. Ε, και ίσως θα πρέπει να το συνδέσουμε αυτό με τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. Ε, θα παρακαλούσα ε, λοιπόν να ε, αυξήσουμε τις απαιτήσεις από 7% των οικολογικών εκτάσεων να το αυξήσουμε αυτό σε 10%. Εάν λοιπόν έχουμε οικολογική αγρανάπαυση, ε, ε, μήπως ο, ο, ε, θα μπορούσε να αποκτεί κίνητρο ε, ότι αν συλλέξει όλα τα στοιχεία και κάνει κάτι θετικό για το κλίμα, θα επωφεληθεί και εκείνος προσεκτικά, θα ε, ε, ε, προσωπικά θα πρέπει να φροντίσουμε να γίνει αυτό. Ευχαριστώ Πετελής, ο Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η δράση για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές τελικά απαιτεί ε, ε, συντήρηση και προστασία του ξύλου και του δάσους. Έχουμε περιόδους ξηρασίας πολύ μεγάλες και έτσι αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύουμε το δάσος, να κάνουμε τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και να εξαλείφουμε την πυκνότητά του, να καθαρίζουμε δηλαδή τις εκτάσεις γύρω από τα δέντρα, ούτω ώστε ο αντίκτυπος της πυρκαγιάς να είναι πολύ μικρότερος. Λοιπόν, τρει τόνοι ένα εκτάριο βιομάζας ε, ξηράς. Ε, πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα όμως να επενθυμίσω ότι καταπολεμήσαμε πολεμήσαμε μάχες σημαντικές θα έλεγα όσον αφορά τους, τους GMS, τους, ε, τους συστοιχεία δωρητόρων, Global Monitoring for Environment and Security. Αυτοί οι δορυφόροι έχουν μέσα ε, τηλεμέτρησης εξαιρετικά αποτελεσματικά και συνεπώς θα μπορούσαμε να ανεκοδομήσουμε ε, τους πίνακες εκείνων ε, των πηγών εκπομπής ε, του άνθρακος και να δούμε ποιες είναι οι περιοχές αυτές που εκπέμπουν περισσότερο. Θα μπορούσαμε συνεπώς να ανοικοδομήσουμε το, να δούμε πού είναι, υπάρχουν συγκεντρώσεις όλων των αερίων του θερμοκηπίου και θα μπορούσαμε έτσι να ε, θεωρήσουμε την αξιόπιστη αυτέ τις μετρήσεις που συμπεριλαμβάνουν και την υγρασία του εδάφους, τη δραστηριότητα την φυτική ε, των καλλιεργών, κυρίως των δασών. Κατά κάποιο τρόπο όλα τα στοιχεία, τα σημαντικά, για αυτό το τομέα να τα διαθέτουμε και μπορούν να δίνονται αυτόματα από τους δορυφόρους, τους GMS και μπορούν να έχουν επιτόπια μέτρηση επίσης, δυνατότητα επιτόπιας μέτρησης, που αυτές οι μετρήσεις οι τοπικές θα μπορούσαν να συμπληρώνουν τα δορυφορικά στοιχεία. Περιμένω να υπάρξει μια δυνατότητα να έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, λεπτομερείς πληροφορίες, χωρίς να δημιουργήσουμε προβλήματα στους γεωργούς που έχουν τις δουλειές τους να κάνουν και έχουν ήδη ακόμα πολλά προβλήματα. Και μπορούμε να έχουμε επιβεβαιώσεις ενός τρόπου, δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε τις μετρήσεις που έρχονται στους δορυφόρους που είναι πολύ αξιόπιστες. Ευχαριστώ. Δεν θα προσθέσω πολλά πράγματα σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν από τον ίδιο τον εισηγητή, τον οποίο τον συγχαίρω για το σχέδιο εκθέσεω του και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Μπάς, ε, όσον αφορά τους ορισμούς και το άρθρο 2, από πλευράς του εισηγητού δεν βλέπω να υπάρχει πρόταση ε, τροποποίησης διευκρινιστική όσον αφορά τη λέξη δάσος Άρα υπάρχουν ε, αντίθετα αυτό το θέμα, όμως θεωρώ ότι ο ορισμός που έχουμε είναι ταυτόχρονα γεωμετρικός και φιλικός προς τη φύση αν θέλετε, αλλά δεν, είναι αρκετά, δεν έχει αρκετά κλιματολογικά χαρακτηριστικά. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο η οπτική άποψη του δάσους ή τι είναι λιγότερο φουντοτό ή τι είναι πραγματικό δάσος, αλλά αν είναι νέο, λίγο πολύ νέο το δάσος ή αν εκπέμπει ή δεν εκπέμπει τα αέρια του θερμοκηπίου. Μήπως θα έπρεπε να φανταστούμε κάποια τροποποίηση που λαμβάνει υπόψη την ηλικία του δάσους και όχι απλώς ε, την γεωμετρία του και επειδή είναι αυτό ο στόχος να λαμβάνει υπόψη κατά πόσο είναι πηγή, άνθρακος ε, ή απορροφά. Γεωμετρικά μπορεί να έχει την ίδια πυκνότητα με δέντρα κάτω των 5 μέτρων κλπ. ή πάνω από 5 μέτρα. Ταυτόχρονα πρέπει να δούμε από πλευράς κλιματολογικής τι γίνεται με τι εκπομπέ. Εκτός αν την ετοιμάσω εγώ ο ίδιος, θα έλεγα να ετοιμάσουμε μια τροπολογία με περισσότερο κλιματολογική χρειά όσον αφορά το άρθρο 2 σημείο Q λατινικό που αφορά τον ορισμό της λέξης δάσος. Για εκείνους Στο τέλος λοιπόν οι Ρώσοι καταφθάνουν στην ΚΟΠ και λένε ότι εμείς έχουμε σημαντικές εκτάσεις δασικές που είναι μονάδες απορρόφησης ε, άνθρακας ε, και ζητάμε συνεπώς πίστοση κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια τόνους ε, άνθρακα διότι είναι πάρα πολύ άδικο αυτό που μας προτείνει η ΚΟΠ. Ευχαριστώ Ευκοσέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν. Θέλω να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, για να αναφερθεί στα σχόλια ή τυχόν αν έχει ερωτήσει, κλπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Αναφέρατε στην αρχή ότι το Λουλουσεφ είναι αρκετά περίπλοκο ακρόνιμιο. Εγώ θα πρότεινα δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το εφήβρε, Πρόκειται περί χαρτοφυλακίου που συζητήθηκε στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα επί σειρά ετών. Έχουμε την απόφαση του Durban και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τα του Durban σε νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στο πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα, αυτός ο τομέας και οι λογιστικοί κανόνες για τον τομέα δεν συμπεριελήφθησαν ε, διότι αναγνωρίσαμε σαφώς ότι ο τομέας αυτός έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προσπαθούμε τώρα να δώσουμε προτάσεις. Δώσαμε μια πρόταση η οποία πιστεύουμε ότι είναι συνετή, ισορροπημένη, λαμβάνω σε υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα. Υπάρχουν πράγματι τα στοιχεία που αποτελούν το βασικό σκοπό της προτάσεως τα απορίσματα του τέρμα να εσωματωθούν σε νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν μία-δύο παρεκκλήσεις που οφείλονται στο ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ασφάλεια δικαίου και ξεκάθαρους κανόνες όσον αφορά το κείμενο που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη σε μία-δύο πτυχές θέλουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι ούτως ώστε τα λογιστικά για τις γεωρικές δραστηριότητες να γίνουν υποχρεωτικά. Ε, έχουμε τα στοιχεία. Ήδη ξεκίνησε η συλλογή των στοιχείων σε όλα τα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια αυτή της περίοδου για το πρωτόκολλο του Κιώτο. Έχουμε στοιχεία επί των οποίων μπορούμε να βασιστούμε και να τα βελτιώσουμε και να βελτιώσουμε τη διαθεσιμότητά τους. Αυτό θα επιφέρει ωφέλη και για τους ε, γεωργούς, διότι τώρα σύμφωνα με αυτά που έχουμε συμπεριλάβει στο λογιστικό σύστημα για τις εκπομπές Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι αρνητικές εκπομπές που συνδέονται με τη γεωργία, μεθάνιο, οξύδιο του νατρίου κλπ. Δεν λαμβάνουν όμως τα θετικά. Διαχείριση των βοσκοτόπων ε, μέσω των γαλακτοφόρων αγελάδων δημιουργεί και θετικά και στοιχεία πίστοσης αν θέλετε, συν ε, που θα μετρηθούν στο μέλλον μέσω της προτάσεως Λουλουσέφ αλλά θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν συμπεριλαμβάνουμε καινούργιο διοικητικό άχθος για τον κάθε γεωργό ούτε για τον δασοκόμο. Είναι υπολογισμοί που γίνονται σε επίπεδο κρατών μελών, ούτως ώστε να καταστεί διαδικασία πλέον διαφανής. Τι γίνεται στον τομέα Λουλουσεφ για την αλλαγή στον τομέα της χρήσεως γεών και της δασοκομείας. Στα περισσότερα κράτη-μέλη, όπως ανέφερα, αυτός ο τομέας παράγει περισσότερο θετικά πίστοση παρά χρέος και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε σύγκριση με πολλούς άλλους τομείς που έχουν συμπεριληφθεί στην ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα. Έχουμε λοιπόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σε κάποιους τομείς δεν γνωρίζουμε αρκετά καλά ποιες είναι οι τάσεις στο συγκεκριμένο τομέα και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σαν μια πολύ συνετή προσεκτική προσέγγιση πρώτα να εστιαστούμε επιλογιστικών κανόνων και μόνο όταν υπάρχουν αυτοί και έχουμε βελτιώσει και εναρμονίσει τον τρόπο υποβολής των πληροφοριών και τους λογιστικούς κανόνες, μετά συζητούμε τον καθορισμό των στόχων. Κατά την άποψή μας, αυτή είναι πολύ προσεκτική και ισορροπημένη προσέγγιση και τα σχέδια δράσης βασικά είναι τα μόνα μέσα μέσω των οποίων μπορούμε να διαμορφώσουμε την πολιτική μας μέσω εγγράφου στρατηγικής το οποίο δεν θέλει να παρέμβει στις εθνικές πολιτικές δασοκομείες αλλά αφορά τις συνέπειες που έχει για το κλίμα το δάσος και πιστεύουμε ότι τα εθνικά σχέδια δράσεως του Λούλουσεφ θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να καλύψουμε κενά γνωστικά. Αν έχουμε εναρμονισμένη προσέγγιση για τη συλλογή των πληροφοριών με στατηγικό τρόπο που προσλέπει στο μέλλον σε όλα τα κράτη-μέλη, τότε γνωρίζουμε καλύτερα το τι συμβαίνει στους τομείς αυτούς στα κράτη-μέλη. Και αυτό αποτελεί καλύτερη βάση για μεταγενέστερη συζήτηση που θα αφορά καθορισμό στόχων. Εκ νέου λέγω ότι η πρόταση δεν δημιουργεί αυξημένη γραφειοκρατία για τους γεωργούς, δεν έρχεται πολύ πρόημα, διότι συζητήθηκε στις διεθνείς συζητήσεις για το κλίμα επί μακρόν και γι' αυτό Πιστεύουμε ότι η πρόταση που κάναμε είναι αρκετά ισορροπημένη, είναι καλή η προσέγγιση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν. Πρωτού να δώσω πάλι το λόγο στον Κρήτον Αρσένη, να πω ότι άσχετα από την αξιολόγηση της έκθεσης αυτής, ε, συνήθως στο Κοινοβούλιο έχουμε δύο αναγνώσεις. Αυτή είναι η κανονική διαδικασία. Κάποιος που διαφωνεί. Μάλλον, εάν υπάρχει συμφωνία, μπορεί να ε, έχουμε μία ανάγνωση, αλλά η κανονική διαδικασία είναι δύο αναγνώσεις. και έχοντας ακούσει τις ε, παρεμβάσεις ε, νομίζω ότι απέχουμε πολύ από συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση όπως ε, και στην Τόχα απέχουμε από συμφωνία αλλά θα ήθελα να το πω αυτό σε όλους και για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και για ε, άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Η διαδικασία σε δύο αναγνώσεις είναι μια διαφανής διαδικασία και όπου μπορεί κανείς ε, να δει σαφώς τα, μπορεί να εξηγήσει κανείς σαφέστερα τα πλεονεκτήματα ενός νομοθετήματος. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να προωθήσετε το θέμα, να προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά σας παρακαλώ να το λάβετε και αυτό υπόψη. Κλείνοντα, να δώσω το λόγο στον ε, εισηγητή, τον Κρήτον Αρσένη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστέψτε με, όχι μία και δύο αναγνώσεις, αλλά ακόμα και συνδιαλλαγή αν χρειαστεί. Τώρα, ε, τα σχέδια δράσης, το μεγάλο ζήτημα που αναφέρθηκε εδώ. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι θέμα διαφορετικών ερμηνεών στο κείμενο. Αν το πρόβλημα είναι η διατύπωση, σίγουρα θα βρούμε κάποιο συμπέρασμα, σίγουρα ε, θα συμφωνήσουμε. Ρωτώ όμως, αμφισβητεί κάποιος εδώ το δικαίωμα και την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βοηθήσει στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. γιατί αυτή είναι και η ουσία αυτή της παραγράφου. Ω προ τα επίπεδα αναφοράς, που νομίζω ότι είναι το δεύτερο θέμα μεγάλης ανησυχίας, ε, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει τις ε, συμφωνίες και τις ε, συζητήσεις για τη διάσκεψη για τις κλιματικές μεταβολές του ΟΗΕ στην Τόχα, γνωρίζουν όλοι ότι κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τα επίπεδα από μόνος του. Μιλούμε για τεχνικές διορθώσεις προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερα, μεγαλύτερη συνοχή. Κανείς όμως δεν μπορεί να αλλάξει το επίπεδο αναφοράς αυτό καθ' αυτό. Τώρα, ως προς το να καταστεί υποχρεωτική η λογιστική καταχώρηση όλων αυτών τα οποία υποχρεωτικώς ήδη πρέπει να αναφέρουμε και αναφέρομαι εδώ και στους βοσκότοπους και στους υγρότοπους στρέφομαι προς τον κύριο Φλόρενς για να σας πω κύριε Φλόρενς ότι ξέρω ότι θέλετε ε, να βοηθήσετε τους αγρότες σας ενδιαφέρουν τα δάση έχετε μάλιστα και δικό σας ε, δάσος και ξέρετε πόσες ε, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι υλοτόμοι στην Ευρώπη και γι' αυτό και θέλετε να τους επειρασπιστείτε και το κατανοώ απολύτως. Ωστόσο, εδώ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ενδεχομένως θέλουν να κάνουν οι αγρότες και λοιποί. Έτσι το ερμηνεύω εγώ, αλλά είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε συζήτηση. Εδώ ε, ε, στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε την κεντρική γραφειοκρατική διαδικασία και δεν μιλούμε καν και για το κτηματολόγιο, θέλετε, ή το μητρό. Όταν ε, όταν αναφερόμαστε στη διαχείριση όλων αυτών των εκτάσεων, ουσιαστικά έχουμε στο μυαλό μας την κοινή γεωργική πολιτική. Δηλαδή, κάτι το οποίο επιδοτείται είναι διαθέσιμο και γίνεται αναφορά για αυτό το πράγμα. υπάρχουν θέματα για τα οποία είναι υποχρεωτική η υποβολή αναφοράς ε, και γι' αυτά ενδεχομένως θέλουμε να έχουμε και υποχρεωτικό χαρακτήρα στη λογιστική καταχώρηση. Η πρόταση λέει ότι θα έχουμε λογιστική καταχώρηση υποχρεωτικά μέχρι το 2020. Δηλαδή σε 8 χρόνια πρέπει να, αποκαλύψουμε, να αποκαλύψουμε τα στοιχεία αυτά. Μέχρι τότε θα είναι στο πλαίσιο εσωτερικής διαδικασίας. Εάν τώρα δεν το κάνουμε αυτό, τι θα συμβεί το εξής α, απλό θα υπολογίζουμε τις εκπομπές Λούλου Σεφ έναντι των στόχων μας και δεν θα τους πιάνουμε τους στόχους αυτούς. Πολλά κράτη-μέλη δεν θα έχουν εξασκηθεί στην απαραίτητη μεθοδολογία και αυτό θα στοιχήσει χρήματα. Ορισμένες χώρες θα είναι έτοιμες να υπολογίζουν τις εκπομπές τους σωστά, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπομπές από την αλλαγή στη χρήση γης, από την αποδάσωση ε, και ούτω καθεξής και να, μπορούν, να μπορεί να γίνεται σωστή αποτίμηση αυτών έναντι των στόχων, άρα θα μειώνουν το επίπεδο των υποχρεώσεών τους για μείωση βιομηχανικών εκπομπών, ενώ άλλες χώρες δεν θα είναι σε θέση να κάνουν αυτό το εγχείρημα σωστά και τελικά πιθανόν να μειώνουν λιγότερο ή μάλλον περισσότερο διορθώνει ο μιλητής ε, να μειώνουν περισσότερο τις εκοπές τους από τη βιομηχανία από ό,τι θα καλούνταν και θα υποχρεούνταν αν είχαν υιοθετήσει τη μεθοδολογία για τη λογιστική καταχώρηση για τις χρήσεις γης και το καθεξής. Σε 8 χρόνια από τώρα θα βρισκόμαστε στην ίδια θέση εδώ, στην ίδια αίθουσα και θα συζητούμε για το ποια χώρα έχει κάνει σωστά ε, τη δουλειά της. Ε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το σωστό εδώ γιατί είναι θέμα χρημάτων και σίγουρα θα παραπονεθούμε και θα γκρινιάξουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Κρήτονα. Τον Ιανουάριο του 2013 μάλλον θα πάμε στην ε, Ολομέλεια, θα έχουμε την ε, πρώτη ανάγνωση. Θα δούμε πότε θα γίνει η δεύτερη. 18 ε, Ιουλίου είναι η προθεσμία για την υπολογή τροπολογιών και στις 19 Σεπτεμβρίου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες στην Επιτροπή Γεωργία. Ε, θα γίνει ψηφοφορία 17-18 Σεπτεμβρίου και στη δική μας Επιτροπή στις 10 Οκτωβρίου. Έτσι ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και φτάνουμε στο επόμενο, το θέμα 6 της ε, ημερήσιας διάταξης. Ε, η Υπουργός Οικονομικών μας, η Γιούτα Χάουκ, μου έχει δώσει το πράσινο φως να συζητήσουμε μαζί τα επόμενα δύο θέματα διότι θέλω να ξεκινήσουμε ακριβώς στις 8, το σημείο 8 στην ημερησία διάταξη. Έχουμε λοιπόν τον Γενικό Προϋπολογισμό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013 όλα τα τμήματα, καθώς και το Πολιτές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020. Ε, ξέρω ότι θα γίνει ε, σημαντική συζήτηση. Ο Βιτόριο Πρόντι ήδη αναφέρθηκε ε, στο θέμα αυτό. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία επί χρόνια ε, υποχρηματοδοτούνται και τίθεται το θέμα εάν ε, θέλουμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Δίνω λοιπόν το λόγο πρώτα στην Ιούτα Χάουγκ για να μας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Να μας παρουσιάσει και τα δύο θέματα της ημερησίας διάταξης. Η Ιούτα Χάουγκ. Ε, συμφώνησα να ε, αναφερθώ στον προϋπολογισμό του 2013, αλλά θα έρθει η εισηγήτρια και Εκεί θα ήθελα να είμαι σκιώδη εισηγήτρια των σοσιαλδημοκρατών, αλλά πασεπτό δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Ε, να αναφερθώ λοιπόν πρώτα στον προπολογισμό του 2013. Ο προπολογισμό ε, δυστυχώ ε, αποτελεί νομοθεσία που αποφασίζεται με μία ανάγνωση. Ε, εγώ το βρίσκω αυτό πολύ δυσάρεστο. Εγώ θα ήθελα δύο αναγνώσει. Ο προπολογισμό του 2013 είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός ε, στην ε, παρούσα ε, δημοσιονομική περίοδο. Τέλη Απριλίου η Κομισιόν προβλέπει 2% αύξηση στις πιστώσει υποχρεώσεων και 6,8% στις πιστώσεις πληρωμών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για ε, το τελευταίο έτος ε, της παρούσας ε, δημοσιονομικής περίοδου και όλα τα προγράμματα στο Περιφερειακό Ταμείο, στο Διασταδιοφωτικά Ταμεία, στον τομέα των ερευνών, είναι πια όριμα να χρηματοδοτηθούν. Η Επιτροπή Προϋπολογισμού του, του Συμβουλίου έχει υποβάλει σχέδιο για ε, το, το Συμβούλιο που θα συναντηθεί μεθαύριο, όπου Ε, προβλέπουν άλλα πράγματα 1,27% ε, αύξηση για τις ε, πιστώσεις υποχρεών και τον, για τις πιστώσεις πληρωμών αύξηση 2,7% κάτι το οποίο είναι γελίο. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό δεν αρκεί καθόλου. Και Καλά είμαι βέβαιη ότι όλοι οι συναδελφοί έχουν διαβάσει τα 15 άρθρα μου, δεν χρειάζεται να τα διαβάσω, αλλά θα ήθελα να πω ότι και όσον αφορά εμάς, εμάς δηλαδή την Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα έχουμε σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά τους οργανισμούς μας. Να σας θυμίσω ότι η Κομισιόν για όλα τα θεσμικά όργανα προβλέπει από το 2013 έως το 2017 ε, να μειωθεί κατά 5% ο προϋπολογισμός. Αυτό σημαίνει ε, κάθε χρόνο 1% ε, λιγότερα. Αυτό το έχει υποβάλει ήδη και στην πρόταση για ε, τους οργανισμούς, τα οποία σημαίνει ότι στην πρόταση του, της Κομισιόν ήδη οι οργανισμοί λαμβάνουν ε, λιγότερα, αλλά αυτό δεν έχει αποτρέψει την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Συμβουλίου να μειώσει ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό. Και μείον 1% όχι όσον αφορά τους πόρους, αλλά και όσον αφορά τη στελέχωση. Για παράδειγμα, ο Οργανισμός Περιβάλλοντος, η ΕΦΣΑ και η ECDC ε, θα έχουν κάθε φορά 1% λιγότερους, λιγότερους σπόρους και 1% λιγότερο προσωπικό. Όσον αφορά την αίμα, είπαν ότι ναι, υπάρχουν μεν νέες ε, αρμοδιότητες, αλλά το μισό των νέων θέσεων ε, διαγράφεται και 1% λιγότερο, λιγότερους σπόρους. Όσον αφορά την ΕΧΑ, την χημικών προϊόντων ε, που θα πρέπει να ε, αξιολογεί και ε, τα φυτοφάρμακα και θα πρέπει να, να δίνει και τις σχετικές άδειε. έχουν μείωση κατά 1% και δεν μιλάω για το 1% της Κομισιόν, ενώ επιπλέον 1% και δεν μπορώ να φανταστώ την κορεπέρ μεθαύριο να τα ανακαλέσει όλα αυτά, παρότι σήμερα στον τριμερή διάλογο κατέστησα σαφές απέναντι στο Συμβούλιο που θα πάμε με όλα αυτά ε, ε, εφόσον υποβάλλουν τέτοιες ανοησίες. Ε, η ΕΓΑ λοιπόν δεν λαμβάνει έγκριση για το 25% των νέων θέσεων. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν έτσι τα πράγματα. Σας το λέω σαφώς. Το ίδιο κάνανε για το πρόγραμμα LIFE, 50% λιγότερο, το πρόγραμμα δράσης για την υγεία 18.000 αλλά ούτως ή άλλως ε, λίγα προγράμματα έχουμε και ε, 18.000 λιγότερα ε, ευρώ. 1,5 εκατομμύριο λιγότερα ευρώ, ευρώ πλοβρέπονται. Δεν αρκούν αυτά και θα πρέπει να περιμένουμε σημαντικές αντιθέσεις και πιθανότατα να μην καταλήξουμε σε προϋπολογισμό τον ε, Δεκέμβριο. Αλλά ναι, αυτό είναι καλύτερο νομίζω και ε, τότε θα ισχύ, ε, ισχύσει η συνθήκη, το οποίο τους άλλους μας δίνει περισσότερα χρήματα στα χέρια μας από αυτό που προτείνει το Συμβούλιο. Έχουμε προπαρασκευαστικές δράσεις και πιλωτικά έργα, τα οποία τα έχουμε υποβάλει στην Κομισιόν για έγκριση. Σήμερα το απόγευμα ε, δεν ε, μπορούσα να ε, να δω την αξιολόγηση της Κομισιόν, διότι ήμουνα στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Αλλά η Γραμματεία, η Εμίλια, έχει στείλει σε όλους την αξιολόγηση αυτή. Όποιο λοιπόν ενδιαφέρεται για τι προπαρασκευαστικέ δράσει και τα ε, πιλωτικά προγράμματα μπορεί να τα κοιτάξει. Υπάρχει λοιπόν εδώ ε, η ιεράρχηση κατά προτεραιότητα των ε, προγραμμάτων, αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Κλείνοντας, τροπολογία για τη γνωμοδότηση, τροπολογίες για τον προϋπολογισμό τροπολογίες για τα ε, πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. 13 ε, Ιουλίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες αυτές ε, και στις 6 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε την γνωμοδότηση. Τελεία. Και θα, θα πάρει το λόγο τώρα η συνάδελφος για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο η συνάδελφο Γιούτα Χάουκ ε, έκανε τη δικιά μου δουλειά, διότι ήδη ανακοίνωσε τι προθεσμίε. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στην συνάδελφο Ματίας, που είναι η Γενική Εισηγήτρια. Κατόπιν, Έχουμε τον ε, συνάδελφό σας, ε, Μανουέλ και την Τάκμα Ροτ Πέρεντ και κλείνουμε και ο Μπάς Άιχαουτ. Ε, κλείνουμε και τον κατάλογο των ομιλητών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι χαίρομαι που είμαι πίσω εδώ, ακόμα και έτσι σύντομα και θα συναντηθούμε ξανά. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια από τα σημεία όπου προσπάθησα να τα εντάξω όλα αυτά, να τα συμπεριλάβω αυτά στην γνωμοδότηση και θα ήθελα να αναφερθώ σε όσα μας είπε η συνάδελφος μου μόλις τώρα όσον αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την γνωμοδότησή μου περιστράφησαν γύρω από το γεγονός ότι συζητάμε για τομείς που είναι υποχρηματοδοτούμενοι. Είναι χρόνια ασθένεια θα έλεγα αυτή. Συνεχώς αποσύρονται χρήματα από αυτά τα προγράμματα που είναι ζωτική σημασία τουλάχιστον κατά την άποψή μου. Καταλαβαίνω ότι κάθε επιτροπή πιθανότατα να πει τα ίδια πράγματα για προγράμματα που εμπίπτουν στην εντολή τους, αλλά πιστεύω ότι αυτά τα προγράμματα είναι ζωτική σημασία. Βλέποντας αυτά που έχουμε μπροστά μας σήμερα, το LIFE, το Health for Growth, και ο μηχανισμός για την πολιτική προστασία της Ένωσης. Ε, αναφερόμαστε σε τα τρία προγράμματα, θέλω να πω κάποια πράγματα. Θα διάβασαν τη γνωμοδότηση κάποιοι συνάδελφοι, είμαι σίγουρη ότι τη διάβασαν, δεν θα διατρέξω όλο το κείμενο. Θα αναφερθώ όμως σε στοιχεία που είναι τα σημαντικότερα για τη σημερινή συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, η μη χρήση της οικονομικής κρίσης σαν δικαιολογία για την μείωση επενδύσεων από τον τομέα των δράσεων για την αλλαγή του κλίματος. Αυτό το θέμα είναι αρκετά σημαντικό για να αποφευθούν υπερβολικές περικοπές. Και γι' αυτό έκανα κάποιες προτάσεις στις παραγράφους 1 και 2 και το ίδιο ισχύει σε όσα σχετίζονται με την αποδοτικότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα ε, και την ε, εμπλοκή σε αυτή την προσπάθεια των μικρομεσών επιχειρήσεων. Υπάρχει ένα φάσμα θεμάτων που είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. επιδιώκοντας το συμπεφωνημένο μοντέλο ανάπτυξης. Ε, όσον αφορά την παράγραφο 3, δεν είμαι σίγουρη που έχουν καταλήξει τα διάφορα κείμενα. Η αρχική πρόταση όμως ήταν ότι θα πρέπει να ξαναδιαθέσουμε πόρους που θα διατεθούν στο Ταμείο για την Παγκόσμια Ποικιλότητα. Στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό ήταν κάτι που είχε αφαιρεθεί από τι δημοσιονομικέ προπτικέ και δεν είχε διατεθεί συγκεκριμένο κονδύλι. Απλώ μία αναφορά γίνεται στι διάφορε στήλε των πινάκων. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συμπεριληφθεί εκ νέου στι δημοσιονομικέ προοπτικέ και με συγκεκριμένο προπολογισμό. Και για το πρόγραμμα Health for Growth αυτό είναι κρίσιμη σημασία υγεία για την ανάπτυξη, πολύ σημαντικό για το κοινό. 10% το ΕΠ καταναλώνεται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και αφορά και το 10% των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να παραμείνουν οι αρχικές ε, χρηματοδοτήσεις, τα αρχικά ποσά. Γνωρίζουμε, το 2020, θα υπάρχει έλλειψη προσωπικού στον τομέα της υγείας. Θα λείπουν περίπου ένα εκατομμύριο άτομα από το απαιτούμενο προσωπικό στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Τώρα που περνάμε μια κρίση μεγάλη, θα πρέπει να υπερασπιστούμε το σημαντικότατο τομέα. Αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας και για την προστασία της δημόσιας υγείας. Και γι' αυτό το υπογραμμίζω όλος ιδιαίτερος αυτό. Τέλος, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέση που υιοθέτησα αντικατοπτρίζει το ότι είναι μία από τις υποσχέσεις που συνεχώς αναβάλλεται στον αφορά τις επενδύσεις. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές δεν έχουν συγκεκριμένο χώρο και χρόνο που συμβαίνουν, άρα θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς πόροι για να καλύπτονται οι ανάγκες που δημιουργούνται όταν συμβούν αυτά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερα εργαλεία, καλύτερα μέσα από αυτά που έχουμε τώρα, τα οποία δεν ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες που υπάρχουν. Στην παράγραφο 8 Ίσως να μην είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Ίσως δεν το διατύπωσα πολύ ξεκάθαρα. Στην παράγραφο 8 λέω ότι πρέπει να διαθέτουμε ένα, ένα ποσοστό 70% για δράση εντός της ε, νόσος και το άλλο 30% για συνεργασία για δράσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεω και νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει και την πολιτική τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ότι θέλουμε να διατηρήσουμε για την εξωτερική συνεργασία ένα επαρκές ποσό. Ο κύριος Φερνάνδης, Χωσέ Μανουέλ Φερνάνδης. δύο λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ ε, τις ξεκινώντα ξεκινώντας από τη Γιούτα Χάουγκ. Θέλω να τη συγχαρώ, ε, έξοχη δουλειά που έκανε, Πολύ καλό το έγγραφο που ετοίμασε. Το έχουμε συνηθίσει να παράγει τόσο ποιοτικά προϊόντα. Να υπογραμμίσω το εξή, ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου το 1% του ΑΕΠ. Αλλά από το 2004 μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από 15 κράτη-μέλη σε 27 κράτη-μέλη. Έχουμε και την ένταξη της ε, Κροατίας επιθύρες έχουμε νέες εξουσίες εμείς και παρόλα αυτά δεν έχω δει κανένα κάτος μέλος να έχει τέτοιες επιδόσεις. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αφορά 94% για επενδύσεις και μόνο 6% του προϋπολογισμού πάει στις διοικητικές δαπάνες ε, και ε, λειτουργικό κόστος. Εμείς θέλουμε νομοθετική αριστεία στις προσπάθειες που κάνουμε Θέλουμε πολύ ποιοτική νομοθεσία, αλλά αν δεν διαθέσει επαρκείς πόρους, ε, τελικά θα χάσουν οι πολίτες μας. Τώρα για τον προϋπολογισμό για το 2013. Το Συμβούλιο εξακολουθεί να ακολουθεί τις προσεγγίσεις που είδαμε και το 2011. Τις ίδιες τεχνικές ακολουθεί. Αρνήθηκε τότε διορθωτικό προϋπολογισμό για αναλήψη υποχρεώσεων και 11 δισεκατομμύρια ευρώ παρέμειναν εκκρεμή. Κάποια κράτη-μέλη στο Συμβούλιο κατάφεραν αυτή την προσέγγιση. Τελικά αυτοπυροβολείται με αυτόν τον τρόπο το Συμβούλιο. Θα έλεγα ότι αποτελεί μαζοχισμό του Συμβουλίου αυτή η προσέγγιση. Υπάρχει έλλειψη σεβασμού για τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Να μην λησμονούμε ότι η έγκριση, η έγκριση των δαπανών στο Συμβούλιο πολύ συχνά οδηγεί σε προβλήματα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι οι πληρωμές θα πρέπει να είναι επαρκείς. Αφορούν δεσμεύσεις, ανέλαβε το Συμβούλιο, αφορούν αυτά τα χρήματα δρομολογηθέντα προγράμματα, αφορά το πρόβλημα χρήματα που οφείλονται. Στο έγγραφο της Utah Haug έχω να προτείνω μία τροπολογία που αφορά την παράγραφο 2 που γίνονται κάποιες συστάσεις εκεί για τους περιβαλλοντικούς στόχους που ισχύουν διασυνοριακά και συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν βάσει συγκεκριμένων προγραμμάτων. Εκεί να προσθέσω όχι μόνο βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά βιώσιμη ανάπτυξη ευφυή ανάπτυξη, ανάπτυξη για όλους. Ταιριάζει με το στόχους του 2020, είναι κοινοί προβληματισμοί αυτοί. Θέλουμε ευφυή ανάπτυξη, όχι μόνο βιώσιμη, και ανάπτυξη για όλους. Πέραν αυτού, μπορώ να συμφωνήσω με τα όσα μας λέει Όσον αφορά την γνωμοδότηση της συναδέλφου Μαρία Ματίας, ας μην κολλήσουμε σε ποσοστά. Θα αποδυναμωθεί η θέση μας εάν κολλήσουμε στα ποσοστά. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν λέτε ότι στο live τα 20% των πόρων πηγαίνουν για την κλιματολογική πολιτική, μάλλον 20% του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Εάν επιλέξουμε αυτή την προσέγγιση θα δημιουργήσουμε προβλήματα για μας, άρα οι αδίποτε στοιχεία με συγκεκριμένα ποσοστά πρέπει να αποσυρθούν από την γνωμοδότηση. Για την παράγραφο 8, η διατύπωση δεν είναι η βέλτιστη. Ίσως δεν είναι και τέλειο το κείμενο στα πορτογαλικά. Ε, όμως δεν νομίζω ότι πρέπει να κολλήσουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Το λέω για μία ακόμη φορά αυτό. Χρειάζονται επαρκή πόροι για την ε, μονάδα για πολιτική προστασία. Αλλά δεν μπορούμε να αναφέρουμε συγκεκριμένο ποσό. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ε, ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες μας. Σας ευχαριστώ που τηρήσατε το δίλεπτο. Η Ντάκμα Ροτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να πάρω και τα δύο λεπτά ε, ε, του Πορτογάλου συναδέρφου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι η συγγήτρια για, το, για τον κανονισμό, για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων στον, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Και παίρνω το λόγο εδώ επειδή είμαι βουλευτής εδώ και πολλά χρόνια. Θα ήθελα να ενθαρρύνω την εισηγήτρια να τονίσει στις εκθέσεις της ότι ε, χρειαζόμαστε ε, προσωπικό υψηλής ποιότητας για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους οργανισμούς. Αυτό φαίνεται και από την έκθεση της κυρίας Χάου και από την γνωμοδότηση της κυρίας Ματίας, ε, αλλά θα ήθελα να τονιστεί περισσότερο. Χρειαζόμαστε μια γενική ε, προσέγγιση, χρειαζόμαστε μια τροπολογία που να καθιστά σαφέ ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν από τη μία μεριά ε, όσον αφορά τις ε, λειτουργικές αρμοδιότητες στον τίτλο 5 να ε, κάνουν μεγάλες οικονομίες και ταυτόχρονα να θέλουν οι αρμοδιότητες αυτές να εκτελούνται ε, στα κράτη-μέλη. Αυτό έχει να κάνει με τον τομέα γεωργίας, ε, με τις έρευνες, ε, ακόμα και, με το περιβάλλον, ακόμα και στο περιβάλλον ισχύει αυτό. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε μία σαφή τροπολογία και να λέμε στα κράτη-μέλη ότι τι, θέλεις χρήματα από το Ταμείο Συνοχής, ποιος Ποιος θα εκτελέσει ε, τα έργα αυτά. Ε, παίρνω και τα δύο λεπτά της Πορτογαλίας. Ε, θέλεις να εισραίουν τα, τα, τα χρήματα από τη Γεωργία ή στο πρόγραμμα Life. θα πρέπει να διαθέσεις και το ανάλογο προσωπικό. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό και παρακαλώ όλους ε, παρακαλώ και όσους δεν, δεν είναι πολύ καιρό εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και τους άλλους να ε, μεταφέρουν ε, στο Συμβούλιο και ε, τους συναδέλφους από την Κομισιόν καλό να θυμίσουν ότι υπήρχε, υπήρχε η Κομισιόν Σαντέρη η οποία έπεσε επειδή ε, δεν είχαν το θάρρος ή τη δυνατότητα να πούν ότι ε, έχουμε τις αρμοδιότητες αυτές, αλλά δεν έχουμε ε, το απαραίτητο προσωπικό για να εκτελέσουμε τα, τα καθήκοντά μας αυτά. Εάν λοιπόν δεν τονίσουμε στο Συμβούλιο ότι πρέπει να διατηρήσουμε τις αρμοδιότητες αυτές, πρέπει να θέλουμε να διατηρήσουμε τη γεωγραφική ισορροπία, θα έχουμε τελικά τόσες μειώσεις στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που δεν θα μπορούμε να εκτελέσουμε λέσουμε τα καθήκοντά μα. Ε, θα ήμουν ευγνώμων αν μπορεί αυτό να το εκφράσει η συγγήτρια, αλλά μπορώ και εγώ να υποβάλω σχετική τροπολογία αν δεν γίνεται τελειώσει. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Μπέρεντε, και για το δίλεπτο. Ε, ήταν μια σημαντική συζήτηση. Θα ήθελα να είναι παρόντες περισσότεροι συνάδελφοι, διότι η συζήτηση αυτή έχει να κάνει με την εκτέλεση, κάτι που συζητάμε εδώ και ένα χρόνο. Και επικροτώ το γεγονός ότι η Κυπριακή Προεδρία Το θέμα της ε, χρηματοδότησης ε, των ε, μέτρων για την αλλαγή του κλίματος το έχει θέσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της. Αλλά ξέρουμε ότι μερικές φορές η φιλία δεν πάει πολύ μακριά, αλλά θα πρέπει να αγωνιστούμε για το θέμα αυτό. Μία κρίση αποτελεί άλλωστε και ευκαιρία. Θέλουμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές που, ε, συμφωνούμε, που αποφασίζουμε στη συμφωνία με το Συμβούλιο και γι' αυτό χρειαζόμαστε και προσωπικό και χρήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη ουσία εδώ και θα πρέπει να βρούμε πιο βιώσιμες λύσεις και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν έχουμε μια σωστή προσέγγιση. Όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Life Plus, εγώ είμαι ο παδός του Life Plus. Όταν βλέπω τα, ε, τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στην εκλογική μου περιφέρεια με το πρόγραμμα αυτό, πόσο μάλλον τώρα που έχει συμπεριληφθεί και η πτυχή του κλίματος εδώ και έχει αναβαθμίσει ε, θα πρέπει να προσέξουμε όμως να μην πούνε ότι αν ορίστε αυξήθηκε το μέτρο αυτό, καλύτερα να, να το μειώσουμε πάλι. Δεν επιτρέπεται να συμβεί αυτό. Και όσον αφορά το πρόγραμμα LIFE, μιλάμε για γελίο ποσό σε σχέση με το σύνολο του ε, προϋπολογισμού. Μιλάμε για χιλιοστά, όχι, ε, μιλάμε για τις χιλίες, όχι τις εκατό του, του προϋπολογισμού. Μιλάμε για τόσο μικρά ποσά. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε το LIFE τουλάχιστον υπό τη μορφή αυτή ε, να υλοποιηθεί και να μην ε, μειωθεί περαιτέρω. Ε, όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τις μειώσεις που γίνονται, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τίποτα να χάσει. Καλύτερο είναι να μην υιοθετηθεί ο προϋπολογισμός παρά να υιοθετηθεί προπολογισμό με τον οποίο να μην μπορούμε να δουλέψουμε. Ε, να πούμε στο Συμβούλιο ότι δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Διότι οι κανόνες λένε ότι αν δεν υπάρχει νέος προϋπολογισμός πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας με βάση τον ε, παλιό. Η συνθήκη της Λισαβόνας ε, μας έχει ε, επιβάλει νέε αρμοδιότητε. χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερα λεφτά. Βλέπουμε όμως ένα όριο μειώσεων του προπολογισμού στο Συμβούλιο. Ο Κυπρίος ε, συνάδελφος ε, ήδη είπε ότι κανένα κράτος μέλος και το είπε αυτό και η κυρία Ροτβέρεντ, δεν μπορεί να επιβιώσει κανένα κράτος μέλος αν δεν έχει ισχυρή και ικανή, ικανή διοίκηση. Θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ανεξαρτησία των οργανισμών. Μπορεί βέβαια πάντα να καλεί κανεί εξωτερικού εμπειρογνώμενε, αλλά την ξέρουμε την συζήτηση. Συχνά αμφισβητούνται αυτοί. Ωραία. Ο Μπά Άιχαουτ είναι τελευταίο ομιλητή στο κατάλογο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Θα είμαι πολύ σύντομος. Αν ε, θέλετε το κάνω και αυτό, μιλάω Ολλανδικά. Θα είμαι πολύ σύντομος πάντως. Συμφωνώ είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα Life Plus. Εμείς όμως ως Επιτροπή όταν συντάσσουμε γνωμοδότηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο γενικότερα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το για το οποίο μιλούμε πράγματι συμβάλλει στο 20% του συνολικού πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αν εμείς, η δική μας Επιτροπή, δεν στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το καν ως προς αυτό, ε, θα ήταν όνειδός μας αυτό, ντροπή μας. Μιλώ και για το 40% του πρασινίσματος ε, της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής. Μιλώ και για το κείμενο Καπούλας Δος Σάντος και στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Ως Επιτροπή οθετήσαμε γνωμοδότηση όπου λέμε το 25% των χρημάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη θα πρέπει να πάει στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στις πολιτικές για το κλίμα. Να τα τονίσουμε δηλαδή ότι ως Επιτροπή ε, θα κάνουμε το παν ώστε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο τελικά να είναι πιο πράσινο, να είναι πολύ πιο νομιμοποιημένο ε, και έτσι να αγωνιστούμε εναντίον των κρατών μελών που θέλουν να περικόψουν κατά 100 δις. Όσοι θέλουν βεβαίως να τα περικόψουν, ψάχνουν να βρουν λόγους να το κάνουν ε, και θα πρέπει να βρούμε τρόπο να μην τους δικαιολογήσουμε και να μην βρουν αυτούς τους λόγους για να τα περικόψουν. Νομίζω ότι τα κατάφερα να μιλήσω μέσα στο δίλεπτο που μου δώσατε. Ευχαριστώ. Τέλεια. Νομίζω ότι σε όλες τις συζητήσεις θα πρέπει να θυμίζουμε ότι εάν Θέλουμε περιβαλλοντικά κριτήρια στη γεωργική και την πολιτική και την πολιτική αλληλεία. Ε, δεν θα πρέπει να χάνονται οι πτυχέ αυτέ τη διαπραγματεύσει. Ε, θα πρέπει να το θυμίζουμε αυτό στους ε, Υπουργού Οικονομικών αλλά και στους Υπουργού Περιβάλλοντος Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι στι ότι στις πρωτεύουσε τους ε, έχουν και υπουργού ε, γεωργίας και ε, και ε, Θα πρέπει να είναι γενική επιτυχία, αλλιώς δεν θα έχουν καθόλου επιτυχία σε αυτό που θέλουν να κάνουν. η προθεσμία για την η υποβολή τροπολογιών για την εκνομοδίτηση της κυρίας ε, Ματίας ε, είναι 17 Ιουλίου 12 το μεσημέρι, θα ψηφίσουμε 19 Ενάτου. 27 Ιουλίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες ε, της έκθεσης ΧΑΟΚ και στις 6 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση για το σημαντικό αυτό θέμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό με τον Υπουργό Περιβάλλοντος ε, της ε, Κύπρου. Ε, είναι η σημαντικότερη προτεραιότητά μας. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το χρηματοδότηση. Περνάμε στο σημείο 8 της ημερησίας διάταξη και, καλό, και καλωσορίζω ε, θερμότατα τον Φίλιπ Λόου, Γενικό Διευθυντή ε, της ε, Γενικής Διεύθυνσης για την ε, Ενέργεια και τον έχουμε καλέσει για να συζητήσουμε μαζί του το θέμα του οικολογικού σχεδιασμού. Δεν θα ήθελα να σπατελήσω άλλο χρόνο, σας δίνω κατευθείαν τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω ε, να μην ξεπεράσω τα δύο λεπτά και να είμαι εξαιρετικά ακριβής. Θα γνωρίζετε ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η συζήτηση για την οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα και θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής σας ε, για τη στήριξη που μας προσφέρατε. Το 17 ε, με 20% της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας θα οφείλεται στη βελτίωση των υφιστάμενων μέτρων για τον οικολογικό σχεδιασμό και τις μεταφορές. Και περιμένουμε τώρα να εφαρμοστούν τα μέτρα τα οποία θα μας οδηγήσουν από το 17 στο 20% και τελικά θα μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και το 33% με τα νέα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού. Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάντοτε στήριζε τις δύο αυτές οδηγίες και για τον οικολογικό σχεδιασμό, την αναδιατύπωση που έγινε το 2009 και την οδηγία, την αναδιατύπωση δηλαδή για την σήμανση, την ετικοθεσία, κάτι που ξεκίνησε ήδη από το 2010. Πολύ έγκαιρα δηλαδή ξεκινήσαμε με την εφαρμογή μέτρων. Έχουμε ε, δύο γενικές ε, διευθύνσεις, δύο αρμόδιους επιτρόπους, τους κυρίους Ταγιάννη και Έτιγκερ και περιμένουμε το 2012 και το 2013 να υιοθετηθούν 29 εφαρμοστικοί κανονισμοί και να αναγνωριστούν τρεις εθελοντικές συμφωνίες με τον κλάδο γενικότερα με στόχο το 2020 να φτάσουμε σε εξοικονόμηση ενέργειας ε, της τάξης των 970 τεραβάτ. Είναι φιλόδοξη αυτή η στόχη και θα ήθελα να πω ότι πρέπει να ε, διευρύνουμε ακόμα περισσότερο το πεδίο εφαρμογής, το πεδίο εφαρμογής αυτών των ε, νομοθετικών κειμένων. Και γι' αυτό κάναμε μελέτες αξιολόγησης και το πόρισμα αυτής της μελέτης ε, ε, αναφέρει ότι είναι τόσο μεγάλο το δυναμικό του πεδίου εφαρμογής που δεν μπορούμε να επεκτείνουμε αυτούς τους στόχους και αυτά τα μέτρα ε, για άλλου είδους προϊόντα και όχι τα ενεργειακά. Είναι νωρίς να γίνει κάτι τέτοιο. Καλό θα ήταν σε τρία χρόνια, το 2014 και όχι νωρίτερα, να αξιολογηθεί εκ νέου η οδηγία αυτή και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών για τον οικολογικό ε, σχεδιασμό ομιλώ. Τώρα, ως προς την οδηγία για τη σήμανση, θα πρέπει να γίνει μια διάμεση αναθεώρηση της εφαρμογή της το 2014, διότι αυτό ξεκίνησε το 2010 ε, και να δούμε πού είναι πιο αποτελεσματικό αυτό το σύστημα οικολογικής σήμανσης και ετικέτας. Τώρα θα ήθελα εν συντομία κύριε Πρόεδρε να αναφερθώ στα σχέδια δράσης βάσει των δύο οδηγιών. Πρώτον, ε, το σχέδιο δράσης 2012-2014 σε σχέση με τον οικολογικό σχεδιασμό περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκριθεί το σχέδιο αυτό τον Ιούλιο όπου περιλαμβάνουμε έναν ενδεικτικό κατάλογο ομάδων προϊόντων και να έχουμε εκεί μία βαθμολόγηση, μία αξιολόγηση κατά σειρά αναλόγως με των δυνατοτήτων που έχουν για εξοικονόμηση ενέργειας. Ε, το πιο καινοτόμο στοιχείο του σχεδίου αυτού είναι ότι πέρα από τα ενεργοβόρα προϊόντα θα χρησιμοποιεί, ε, θα αναφέρεται και στα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια, όπως είναι ας πούμε τα υλικά μόνωσης ή τα παράθυρα και τα κουφώματα. Χάρη στη δική σας δέσμευση έχουμε καταφέρει να έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά μπορούμε να καταφέρουμε ακόμα περισσότερο, ε, περισσότερα. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο νομοθετικό έργο αυτό για τον οικολογικό σχεδιασμό και θα έχουμε προπαρασκευαστικές ομάδες. Όπως σας είπα, αναμένουμε να υιοθετηθούν 32 αποφάσεις, 29 εφαρμοστικοί κανονισμοί και 3 επιβεβαιώσεις ε, συμφωνιών εθελούσιου χαρακτήρα και φέτος έχουμε υιοθετήσει ήδη 3 κανονισμούς ε, για τον οικολογικό σχεδιασμό κτλ. και μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουμε υιοθετήσει ακόμα 8 ε, κανονισμούς σχετικούς με το θέμα τελικά θα φτάσουμε σε εξοικονόμηση ενέργειας ε, της τάξης ε, το 450 τεραβάτ και έτσι θα μας μείνει για την επόμενη χρονιά το 2013 ε, να δουλέψουμε για να εγκρίνουμε και άλλους κανονισμούς και άλλες εθελούσεις συμφωνίες για τα υπόλοιπα 530 τεραβάτ που μένει να εξοικονομήσουμε. Ε, για να ολοκληρώσω τη σκιαγράφηση της εικόνας αυτής, θα σας πω ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και τους υφιστάμενους κανονισμούς για ορισμένες ομάδες προϊόντος και εκεί πρέπει να αξιοποιήσουμε, εκεί βρίσκονται οι περισσότερες δυνατότητες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να έχουμε όσο να το μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Και βεβαίως ε, για να γίνει αυτή η δουλειά θα εξαρτώμαστε πολύ από το διάλογο που θα έχουμε με εσάς εδώ στο Κοινοβούλιο για να έχουμε απτά και σωστά και καλά αποτελέσματα. Η εποπτεία της αγοράς, η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά είναι πολύ σημαντική. Βεβαίως ε, κάνουμε διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, με τα, τις ομάδες καταναλωτών, με τα κράτη-μέλη, ε, με όλους τους ενδιαφερομένους και προγραμματίζεται κοινή δράση με το πρόγραμμα ε, για την έξυπνη Ευρώπη ώστε να στηριχθούν δράσεις για την εποπτεία της αγοράς. Και θα ενισχύσουμε την συνεργασία μεταξύ Εθνικών Αρχών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω των ομάδων ad hoc επιτόπου διοικητικής συνεργασίας. Και τέλος, ε, θα ήθελα να σας ευχηστήσω την προσοχή στην ανάγκη αξιοποίησης πολλών πόρων ε, προκειμένου να έχουμε αυτή την νομοθετική δραστηριότητα. Ανακοινώσεις, ε, τυποποίηση, εφαρμογή, υλοποίηση. Θα χρειαστούμε τη βοήθεια του κοινού ερευνητικού κέντρου στην Ευρώπη και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Καινοτομία. Ε, θα στηριχτούμε σε, όλα αυτά, σε όλους αυτούς τους φορείς και έχουμε τις απαντήσεις από τις ομάδες των καταναλωτών ε, για το, την ενεργειακή σήμαση και για τον οικολογικό σχεδιασμό. Ε, μέσω του, ενός διάβλου που έχουμε θεσπίσει στην διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε και ένα help desk που ε, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο επίσης. Έχουμε εσωτερική συνεισφορά ως προς την τυποποίηση, τυποποίηση και θα λάβουμε υπόψη μας όλη αυτή την ε, συνεισφορά εκεί για τις 39 ομάδες προϊόντων. Σίγουρα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν όλα αυτά το 2012 και το 2013. Θα γνωρίζετε τα διάφορα συμφέροντα της βιομηχανίας, θα γνωρίζετε τα, τις απαιτήσει και τις επιθυμίες των καταναλωτών. Μία σχέση κόστους-οφέλειας είναι εξαιρετικά σημαντική. Η επίτευξη σωστής ισορροπίας είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε διεξάγει ευρείες συζητήσεις για πολλές ομάδες προϊόντων. Ε, έχουμε από θέματα όπως οι καφετιέρες και η ενεργειακή τους κατανάλωση που δεν ενδιαφέρει σχεδόν καθόλου μέχρι και θέματα όπου η κατανάλωση των προϊόντων ενδιαφέρει πάρα πολύ όπως είναι οι καυστήρες ε, μεταξύ άλλων. Ε, είναι πολύ σημαντική η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών, πόσο τελικά οδηγούν στην ε, εξοικονόμηση ενέργειας, πόσο ε, προσφέρουν μια καλύτερη σχέση ως κόστους ωφέλειας στον, στους καταναλωτές, στους πολίτες. Περιμένουμε πολύ ζωντανή συζήτηση για κάθε μία από τις ομάδες προϊόντων. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια συζήτηση για τους λέβητες και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σύντομα. Ε, συζητούμε με τους ενδιαφερομένους και περιμένουμε ε, μέχρι το φθινόπωρο να υπάρξουν αποτελέσματα. Ένας δεύτερος γύρος κανονισμών θα ε, υπάρξει σε σχέση με τους λαμπτήρες οικιακής χρήσης και αυτό είναι κάτι στο οποίο τα μέσα μαζικής επικοινωνίας θα στραφούν αμέσως για να ρίξουν φως σε όλη αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να χειριστούμε πολύ σωστά τις ομάδες προϊόντων όπου υπάρχει αίσθηση ότι θα υπάρξει αντιστάθμισμα μεταξύ της τιμής που πληρώνει κανείς για να αποκτήσει αυτό το προϊόν και του ωφέλους τελικά που παίρνει ως καταναλωτής από τη χρήση του. Αυτά προς το παρόν κύριε Πρόεδρε, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φιλιπ Υπάρχουν και κάποια επίμαχα σημεία, τα οποία σίγουρα θα ακούσουμε στην ε, γενική συζήτηση. Πάντως ενδιαφέρον είναι ότι ακούσαμε ότι ε, ο οικολογικός σχεδιασμός δεν αφορά μόνο τον τομέα της ενέργειας. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την έκθεση Ζήμπερ. Υπάρχουν λοιπόν τομεί όπου δεν το φαντάζεται κανεί καν. Είχαμε και την έκθεση iHout σχετικά με την ε, απόδοση των πόρων στην Ευρώπη. Υπάρχουν πόροι τους οποίους θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, και να εκμεταλλευτούν προσεκτικά όπως είναι η ενέργεια αλλά όπως είναι και το νερό. Ε, είναι δύσκολο το θέμα λοιπόν του οικολογικού σχεδιασμού. Θα πρέπει να το μεταφέρουμε με καλό τρόπο λοιπόν στο κοινό και χαίρομαι για αυτό που είσαστε εδώ σήμερα και έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα αυτό μαζί σας. Πέτερλιζε, Κρίς Τέιβις και Μπάς Άιχαουτ έχουν ζητήσει το λόγο. Ξέχασα κάποιον. Αλλιώς θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Αυτοί οι τρεις. Πρώτα ο Πέτερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά. Ε, θα ήθελα Ε, να ανταποδώσω τις ευχαριστίες για τη συνεργασία πάνω στην ε, οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία και με την Γενική Διεύθυνση και με τον κύριο Έτενγερ και το γραφείο του. Ε, για την Επιτροπή μας ήταν πολύ σημαντικό το θέμα της εμπορίας εκπομπών και καταφέραμε να βρούμε μια κοινή λύση υπό τη μορφή μιας δήλωσης της Κομισιόν. Τώρα όμως ανησυχούμε λίγο, διότι νομίζω ότι υπάρχουν ε, κάποιες ενέργειες. Υπάρχει μία έκθεση ε, της ε, Business Europe που λέει «Σας παρακαλούμε, Κομισιόν, αγνοήστε όλα όσα είπε το Κοινοβούλιο». Αυτό όμως δεν γίνεται. Είμαστε θεσμικό όργανο. είχαμε δραστηριότητα λόβια από πλευρά της Business Europe, αλλά επιμείναμε στο θέμα αυτό. Είμαι γιατρός και ε, το βλέπω ως εξής. Ε, η Κομισιόν έκανε μια διάγνωση τον Ιούνιο ε, ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι. Πριν τις διακοπές, λοιπόν, θέλουμε την, την σχετική έκθεση. Αλλιώς δεν μπορεί να υποστηρίζει η Κομισιόν ότι είναι επίγον το θέμα όσον αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό. Είναι κρίμα που μιλάτε εδώ μπροστά σε τόσο λίγους ευρωβουλευτές. Είμαστε η αρμόδια επί της ουσίας ε, έκθεση. Ε, όταν ακούμε τον κόσμο υπάρχουν, αρνητικά, υπάρχουν θετικά, υπάρχουν και αρνητικά θέματα εδώ. Ε, θα πρέπει νομίζω να πάρουμε λοιπόν όλο τον χρόνο που απαιτείται. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό για την ευρωπαϊκή πολιτική και είμαστε εμείς αρμόδιοι επί της ουσίας. Μπορεί να είναι τυπικό το θέμα, αλλά στην, ε, γνωμοδο... στην ε, ημερήσια διάταξη λέει απλά εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Γενικό Διευθυντή όμω είναι. σω θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό στο μέλλον περισσότερο. Αλλά βέβαια είναι μάλλον τυπικό το θέμα. 970 ε, τεροβατόρες ε, αναφέρατε, ε, τις οποίες μπορούμε να εξοικονομήσουμε μόνο με τον οικολογικό σχεδιασμό. Αυτό είναι το σύνολο της παραγωγής των, πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι μέχρι το 2020 θα κλείσουμε όλα τα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη. για τέτοια νούμερα μιλάμε αναφερθήκατε στη θέρμανση, αναφερθήκατε στο νερό. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο μέτρο, διότι θα πρέπει να δούμε πού υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες και τι γίνεται όσον αφορά ε, τις ε, καφετιέρες, τις τοστιέρες ε, και τα τηλέφωνα του ντους. Ε, υπάρχουν πολλά θέματα ε, τα οποία ε, δεν έχουν να κάνουν άμεσα με το, με το σύνολο του πληθυσμού, όπου μπορούμε να κάνουμε εξοικονομήσεις. Υπάρχουν όμως ε, και θέματα που μπορεί να κάνει ο, ο καθένας. υπάρχουν οι λάμπες αλογόνου και άλλες λάμπες που θέλουμε, άλλες λάμπες οικονομίας. Δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε τις λάβες αυτές, να αποσύρουμε τις, λάβες, ε, τις παλιές λάβες ε, ε, από το εμπόριο. Ε, διότι είπαμε ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το αποφασίσει. Θα ήθελα να τονίσω ε, αυτό που είπατε εσείς σχετικά με την ε, εποπτεία της αγοράς. Σημαντικό κομμάτι της οδηγίας αυτής είναι ότι έχει να κάνει και με τις εισαγωγές. Μπορούμε λοιπόν να επιβάλλουμε ένα πρότυπο το οποίο θα εφαρμόζεται και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θέλουν οι τρίτες χώρες να εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει λοιπόν να γίνονται έλεγχοι ώστε να διαπιστώνουμε εάν ε, πράγματι εξοικονομούν ενέργεια τα εισαγόμενα προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να σχεδιαστούν τα ε, ε, μέρους μέτρα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ελέγχονται επίσης. Ο Κρίς Ευχαριστώ Πρόεδρε έχουμε δηλητηριώδη πολιτική συζήτηση για την Ευρώπη στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολύ συχνά αναφέρεται τα μέλη του Κοινοβουλίου αυτού και τα μέλη του Κόμματο Ανεξαρτησία του Ηνωμένου Βασιλείου ότι μπήκαμε στην κοινή αγορά και δεν θέλουμε στου κανόνε. Ήταν απλώ εμπορική σχέση και δεν καταλαβαίνουν ότι η αγορά χρειάζεται κανόνε και ρυθμίσει για να λειτουργεί και δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο κανονισμό, οδηγία, αυτή η περίπτωση από αυτόν. Μου αρέσει αυτό το νομοθέτημα. Είναι ένα νομοθέτημα το οποίο συνεπάγεται αλλαγές που θα μειώσουν το κόστος για τους καταναλωτές. Προωθεί την καινοτομία. Μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της θέρμανσης του πλανήτη και κάνει προτάσει καλύτερη χρήση των πόρων. Και αν το επεκτείνουμε περαιτέρω, πέρα από τα ενεργειακά θέματα και πάμε στο νερό κλπ. κλπ. Άρα είναι ένα υπέροχο, υπέροχο παράδειγμα το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πράγματα που θα κάνουν τη διαφορά. Τι κάνουν οι, τι, τι έκαναν οι, Ρωμα... οι Ρωμαίοι για σας, τι έκανε ας πούμε η Ευρώπη για σας μπορούμε να πούμε αντίστοιχα. Ε, τον οικολογικό σχεδιασμό έχει εισαγάγει. Ε, χαίρομαι που εξήγησε ο Πίτερ Σαφώ αυτά που, που έπρεπε. Έχει διακοπεί το ήχο στο το μικρόφωνο του μιλητού δυστυχώς. Uh, ο Νάιτζελ Φάρατζ με έπιασε, με τσίμπησε. Λοιπόν, χαίρομαι που ο Πίτερ Λίζε εξήγησε σε τι αναλογούν τα 970, 970 ε, τεραβατόρες. Δεν ξέρω αν έχει διαπιστώσει, αν έχουν κλείσει όλοι οι πυρηνικοί σταθμοί στη Γερμανία ή πρόκειται να κλείσουν. Ο κύριος Διευθυντής θα μπορούσε να μας εξηγήσει περαιτέρω το θέμα. Εντάξει, η οδηγία είναι πολύ νέα, αλλά από τις αναφορές που είδα μέχρι τώρα, οι οικονομίες, ε, πολλές οικονομίες θα μπορούσαν να αποδοθούν σε αυτή. Ε, και φαίνονται σαν να είναι απλέ ε, εξοικονομήσει ενέργειας λόγω αποδοτικότητα βελτιωμένης. Όσο περνά ο χρόνος θα κάνει και περισσότερα, θα έχει περισσότερα αποτελέσματα η οδηγία. Το ερώτημά μου είναι, τι περισσότερο μπορούσαμε να πετύχουμε. Αναφέρατε κύριε Διευθυντά ε, το τι αναμένετε. Αλλά δεν ε, αυξήσατε τον πύχη στον αφάσι της Δεν είπατε αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε εάν διαθέταμε περισσότερου πόρου, περισσότερο προσωπικό, αν βρίσκαμε τρόπου για να επιταχύνουμε ε, τη διαδικασία, αν βελτιώναμε την εφαρμογή στην αγορά. Έχω μια έκθεση εδώ, εξασέλιδη από μη κυβερνητικέ οργανώσει με συστάσει που δεν θα σα διαβάσω, αλλά είμαι σίγουρο ότι ε, έχουν ε, απευθυνθεί και σε εσά. Ε, τι δυναμικό υπάρχει, πόσο καλύτερα μπορούσαν τα αποτελέσματα από ό,τι προτείνατε εσεί και τι μπορούμε να κάνουμε για να τα ελοπίσουμε αυτά. Ευχαριστώ, Chris David. Chris Eichert. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τριβήσω και να αναφερθώ όσον αφορά τη σημασία του νομοθετήματος, διότι ήδη ο Πίτερ και ο Κρίστα αναφέρανε αλλά διερωτώμην όταν μιλούσατε για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ κατασκευαστών και καταναλωτών και συνήθως μας αρέσει η ισορροπία, αλλά αυτό το νομοθέτημα είναι υπέρ εκείνου που ε, λειτουργούν πολύ καλά. Και επίτευξη ισορροπίας τι σημαίνει ότι πάμε στο μέσο όρο. Ενώ εδώ αυτό το νομοθέτημα θα έπρεπε να σπρώχνει, να προωθεί εκείνους που ηγούνται μέσω καινοτομίας. Και έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ πράγματι προσπαθεί να εξορροπήσει την κατάσταση με αυτούς που μένουν πίσω. Ε, οι καυστήρες ε, και ε, από ό,τι είπατε μάλλον καλά κάτι γίνεται εκεί. Υπήρχε διαβούλευση πέντε χρόνια από ό,τι ξέρω. Ε, ακόμα και ο ΠΟΕ τελικά αναφέρθηκε κλπ. Αλλά εξακολουθώ να ακούω ότι λέτε ότι προσπαθούμε να πετύχουμε μια ισορροπία το φθινόπωρο. Σας παρακαλώ, μπορείτε να καταφέρετε καλύτερα. Ε, τα συμπεράσματα ήταν σαφέστατα, η πρόταση υπάρχει, τη γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε επίση ότι αυτή την Παρασκευή έγιναν κάποιε συναντήσει με, τη, με εκπροσώπου τη γερμανική βιομηχανία. Αλλά δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει μια πρόταση, θα έπρεπε αύριο ακόμα να υποβληθεί. Αν αυτό είναι πολύ δύσκολο, καλώ αρχέ Σεπτεμβρίου μέσω κατεξοδότηση πράξεω. Περιμένουμε. Είναι τα σημαντικότερα θέματα αυτό και η επίτευξη της ισορροπία έχει γίνει εδώ και πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια γίνεται αυτή η προσπάθεια και ελπίζω να προχωρήσουμε πιο γρήγορα γιατί ήσασταν πολύ αόριστο. Είπατε κάπου το φθινόπωρο. Μετά για την αναθεώρηση είπατε 2014 αλλά υποθέτω ότι πρόκειται περισφάλματος αλλά είναι 2013 και ελπίζω ότι τότε πραγματικά θα ακολουθήσουμε το μοντέλο εκείνων που προχωρούν καλύτερα όπως το έκανε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Γερμανία. Ε, αν μπορείτε να πείτε πάνω σε αυτό κάτι. Ευχαριστώ. Ιάννα Βαϊσκέπα. Ευχαριστώ. Θα είμαι συντομότατη όπως υποσχέθηκα. Θα ήθελα να μιλήσω για αυτά που έθιξε ο Πίτερ Λίζε δεν θέλω απλώ να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Επιτροπή περιβάλλοντα προσπαθεί να το περάσει αυτό, να το περάσει πιο γρήγορα κλπ. Υπάρχουν κάποια κρίσιμα σημεία που περιέχονται, αυτά που ανέφερε προηγουμένω ο Πίτερ Λίζε, προϊόντα τα οποία θα συζητηθούν στο δημόσιο όπω οι καφετιέρες ή όπω οι κεφαλές του ντου κλπ. Στα τηλέφωνα του ντου. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε για του λαμπτήρες στα σπίτια, ε, στι κατοικίε, θέλετε να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό, τι σχεδιάζετε ακριβώ να κάνετε, ποια είναι τα συγκεκριμένα σχέδιά σα. Νομίζω ότι ήταν σφάλμα μα που δεν εξηγήσαμε αυτά τα θέματα στου ε, εκλογεί μα τότε ότι είχαμε νέε τεχνολογίε, ότι νέε τεχνολογίε δημιουργούν νέε δυνατότητε. σω να πιεστήκαμε πολύ και να μεταξηγήσαμε. Οπότε ε, επικρίνω αυτό το σημείο όσον αφορά το φωτισμό στις κατοικίες. Νομίζω ότι χρειάζεται καταρχάς να εφαρμόσουμε τα ήδη συμπεφωνημέντα. Ευχαριστώ την Άνια Βάις Κέρπερ ε, και η Γερμανική Προεδρία τότε είχε αναφερθεί στο θέμα αυτό με την ε, οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό. Σε όλες ε, αυτές τις ε, προτάσεις ε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο οικολογικός σχεδιασμός μπορεί να είναι σε εποχή κρίσης και σε εποχή περιορισμένων πόρων ακρογωνιαίος λίθος και θα πρέπει να το μεταφέρουμε αυτό στον κόσμο. Δεν είναι απαραίτητα φρένο πολύ συχνά πρέπει να εξηγούμε την ε, πολιτική και γι' αυτό είναι πολύ καλή και η προσέγγιση του Γερμανού ε, Υπουργού Περιβάλλοντος. Εάν λοιπόν μπορεί κανείς να ε, εξοικονομήσει το 35% της κατανάλωσης νερού σε ένα νοικοκυριό, αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα. Και η κυρία Ροτμπέρεντ αναφέρθηκε στα προαιρετικά μέτρα, τις προαιρετικές συμφωνίες. Το γνωρίζουμε αυτό από τον τομέα των αυτοκινήτων. Ε, τότε σε μένα χτυπάνε καμπανάκια. Εγώ αρχίζω και φοβάμαι τότε, διότι... Ένα ξέρω, ότι δεν εφαρμόζονται τα προαιρετικά μέτρα. Μήπως μπορείτε να αναφερθείτε και σε αυτό το θέμα, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Χαίρομαι διότι πραγματικά και εγώ και όλο το τμήμα του οποίου ηγούμε θεωρούμε ότι αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Πράγματι πρέπει να ε, είμαστε διεκδικητικοί γιατί έτσι θα βοηθήσουμε όχι μόνο την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της ε, οικονομίας. Ε, μπορεί με να μιλώ ορισμένες φορές συντηρητικά, αυτός είναι και ο βασικός λόγος που σας λέω ότι έχουμε υποβάλει την πρόταση για τους καυστήρες και τους λέβητες και θα συνεχίσουμε να τις υπερασπιζόμαστε τις προτάσεις αυτές. Το πιο σημαντικό είναι να εξηγήσουμε τα ωφέλη ε, σε αυτούς που πρέπει να τα εξηγήσουμε, όπως ζητεί και ο αρμόδιος επίτροπος. Δεν θα τα παρατήσουμε. Έχουμε το σχεδιασμό μας για το 2012 και το 2013 και όντως έχουμε ε, τους λαμπτήρες οικιακής χρήσης, τις ηλεκτρικές κούπες, τις ε, συσκευές που τίθενται σε λειτουργία αναμολή, αναμονής, ε, τις καφετιέρες, πάρα πολλά πράγματα. Μπορώ, ο κατάλογος είναι εξαντλητικός. Καλό θα ήταν να πετύχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε προβλέψει και θα μου άρεσε βεβαίως να είμαι σε θέση να πω ότι με την αναθεώρηση ε, τη υφιστάμενης νομοθεσίας πετυχαίνουμε περισσότερα από το 1% που είναι το ανώτατο των εξοικονομήσεων που προβλέπεται εδώ. Αλλά κάθε δουλειά στον τομέα αυτό περνάει από τρία στάδια. Πρώτον, αξιολογούμε κάποια νέα ομάδα προϊόντος και αν υπάρχει μια προκαταρρετικη σχέση κόστους ωφέλειας εκεί και αναξίζει αξίζει τον κόπο να γίνει έρευνα γι' αυτό. Αυτό κάναμε με τις καφετιέρες και φαίνεται ότι και να εμβαθύνουμε δεν είναι πολλά υποσχόμενο το πεδίο αυτό γιατί εξαρτάται από τη συμπεριφορά του καθενός από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί την καφετιέρα η εξοικονόμηση ενέργειας εκεί. Ε, και βεβαίως πάμε σε πολύ πιο σοβαρούς τομείς όπου η κατανάλωση ενέργειας είναι εξαιρετικά ε, σημαντική στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο ε, για κάθε νοικοκυριό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να είμαστε επιφυλακτικοί και συντηρητικοί αν θέλετε για να είμαστε σίγουροι ότι θα ασχοληθούμε με πεδίο όπου σίγουρα θα πετύχουμε. Αυτό ναι στην αρχή. Από εκεί και πέρα, όταν μπούμε στη μάχη δεν θα ε, αναζητήσουμε ισοπαλία, ούτε αντιστάθμισμα ε, και ανταλλάγματα προς τη βιομηχανία. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε ως προς την αποδοτικότητα, την εξοικονόμηση και τη βελτίωση γενικώ ε, ε, της κατανάλωσης. Ο Επίτροπος Έτιγκερ και όλη η ομάδα που τον υποστηρίζει έχουν πολύ μεγάλες φιλοδοξίες ως προς αυτό. Θα γίνει πολλή δουλειά και ήδη γίνεται για το 2012 και 2013. Άκουσα τη συζήτηση για το πόσο προσωπικό σημαντικό πώς οι ανθρώπινοι πόροι είναι διαθέσιμοι για την εφαρμογή αυτής και άλλων οδηγιών. Ε, θέλω να σας πω ότι αξίζει να επενδύσει κανείς σε ανθρώπους ε, για το στον τομέα αυτό προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα. Ε, οι άνθρωποι της ομάδας μου, οι οποίοι δεν είναι και πάρα πολλοί, πιέζονται αρκετά και κάνουν πραγματικά πολύ σπουδαία δουλειά έχουν ήδη κάνει και κατά τη φάση των διαπραγματεύσεων και θα συνεχίσουν να κάνουν μια δουλειά με πολύ μεγάλη προσοχή ε, στη λεπτομέρεια. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Ε, για να απαντήσω σε εσά, κύριε Πιτελίζε, θα σα πω ότι όντω εγώ ήμουν εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον τριμερή ή τριγωνικό ε, διάλογο και εγώ έλαβα την πρότασή σα για τα μέτρα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση και στη συνέχεια ε, εγκρίθηκε το θέμα από το Σώμα των Επιτρόπων. Όποια και αν είναι τα συμφέροντα δηλαδή της βιομηχανίας ή του κλάδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε υπέρ αυτής της δήλωσης και αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό. Ε, δεν μιλάω βεβαίως ε, εκ μέρους και της Επιτρόπου Κόνι Χέντεγκάρντ, αλλά έχω την εντύπωση ότι το ίδιο πιστεύει. Η πρόταση αναθεώρησης πριν από τις ε, διακοπές τίθεται ένα αμφιβόλο. Ελπίζω ότι θα βοηθήσουν οι φωνές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι είναι πολύ σημαντικό θετικό το σημάδι για μακροπρόθεσμες επενδύσεις που θα δοθεί εάν φανεί ότι ένα σύστημα εκπομπής εμπορίας λοιπόν και δουλεύει σωστά. θα πρέπει να στηρίξουμε τους συναδέλφους μας που εργάζονται στο πεδίο ε, για τις κλιματικές μεταβολές και είναι κάτι που κάνουμε. Και θέλω να πω και το εξής. Αν δείτε τους ξεχωριστούς τομείς και πεδία δράσης, ναι, γίνεται συζήτηση για τα τηλέφωνα του ντους, ε, για, το, για τέτοιου είδους πράγματα κατά πόσο αξίζει τον κόπο δηλαδή να, έχουμε αυτές τις επιδιώξεις και να ε, τα βάλουμε αυτά στο επίκεντρο του σχεδίου δράσης μας. Θα σας πω την άποψή μου. Σε τεχνικό επίπεδο είμαστε πεπισμένοι ότι μπορεί να γίνει ουσιαστική εξοικονόμηση εκεί. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά λέτε, όταν ε, μπαίνουμε σε τέτοιου είδους χωράφια πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ως προς την επικοινωνιακή μας πολιτική, τις ανακοινώσεις που έχουμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και κατά τη διάρκεια της υποβολής των προτάσεων και βεβαίως ε, αυτή τη συζήτηση διεξάγει αυτή τη στιγμή η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κατά πόσο θα συμπεριληφθεί αυτή η ομάδα προϊόντων στο σχέδιο εργασίας. Εμείς πιστεύουμε ότι όντως μπορεί να γίνει εξοικονόμηση και ίσως περισσότερο εκεί από ότι ε, σε άλλα πεδία. Τώρα, ως προς τους λαμπτήρες, πρέπει να δώσουμε πολύ ξεκάθαρες εξηγήσει για το ποιες είναι οι προθέσεις μας και να μην επαναλάβουμε τα λάθη, όχι τα δικά μας, δεν θα έλεγα ότι εμείς έκαναμε λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, τα λάθη τα οποία έκαναν σύσσωμα τα πολιτικά θεσμικά όργανα αλλά και οι εταιρείε οι οποίες ε, λάνσαραν νέα προϊόντα στην αγορά χωρίς να έχουν πραγματική αντίληψη του τρόπου με τον οποίο ε, τα ερμηνεύει και τα αντιλαμβάνεται τελικά ο ίδιος ο καταναλωτής. Ε, θα έχουμε λοιπόν νέες κατηγορίες σε αυτή την ομάδα. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ως προς τις διάφορες κατηγορίες για τους λαμπτήρες. Γιατί ξέρετε, όταν μπαίνει κανείς σε αυτό το χορό των συζητήσεων πρέπει να χορέψει μέχρι τέλους. Θα πρέπει λοιπόν να βγάλουμε σωστή ανακοίνωση ευθύ εξ αρχής για αυτή την ομάδα προϊόντων. Από εκεί και πέρα. Αναγνωρίζω ότι δεν είμαστε επαρκώς ακριβείς στη διατύπωσή μας για τις μελλοντικές δυνατότητες. Πιστεύω όμως ότι η αναθεώρηση των 11 υφιστάμενων κανονισμών πράγματι θα προσφέρει ένα αποτέλεσμα που θα ξεπεράσει κατά πολύ το 1%. Εμείς δημοσίως μιλούμε για 1%, αλλά τελικά εννοούμε τουλάχιστον 1%, εννοείται παραπάνω. Και ως προς τις διαπραγματεύσεις για την οδηγία, για την ενεργειακή αποδοτικότητα, όχι μόνο μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αλλά και με τους εξωτερικούς παράγοντες, ε, η πρόκληση είναι να δημοσιεύσουμε σωστά πόσο ακριβώς θα ε, από την εφαρμογή κάθε ενός έργου. Τώρα, οι 970 τέρα βατόρες ε, είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να σας μεταφράσω σε μεγαβάτ αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, μπορώ να σας πω ότι σίγουρα ε, αυτά που έχουμε ήδη επιτύχει ε, ισοδυναμούν με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης, ισχύω της τάξης των 500 ΜΒ. Το λέω αυτό για να έχετε μια τάξη Το δύσκολο όμως είναι ότι έχουμε ήδη υπολογίσει πολλές από τις εξοικονομήσεις σε αυτή τη βασί, γραμμή βάσης. Μιλούμε για εκατοντάδες ε, σταθμούς ε, ισχύως το της των 500 ΜΒ ή εκατομμύρια ανεμογεννήτριες. Δηλαδή ε, μια τάξη μεγέθους είναι αυτή. Το πόσο θα εξοικονομηθεί. Θα εξοικονομηθεί τόσο όσο θα παρήγαγαν ε, τα στοιχεία που σας είπα, οι σταθμοί που μόλις ανέφερα. Αυτό τι είναι μια σύγκριση, μια μεταφορά που μπορώ να κάνω για να είμαι κάπως πιο εύγλωτος. Είναι, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω σε αυτό το στάδιο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη και για την ενθάρρυνση ε, σας για το ότι συνεχώς μου λέτε να μην ε, υποχωρήσω. Μια ερώτηση μόνο. Ε, ως προς τους καυστήρες, πέντε χρόνια ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, αλλά είπατε πέντε χρόνια χρειάστηκαν για να ε, δοθούν εξηγήσει. Ναι, απαντάει εκπρόσωπος της Επιτροπής, στις αρχές Σεπτεμβρίου περιμένουμε να ληφθεί απόφαση για τους καυστήρες. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε έτσι την συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Φίλιπ Λόου που είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί του το θέμα του οικολογικού σχεδιασμού, την κατάσταση, το τι είναι σχεδιασμένο και όσον αφορά την μετατροπή είναι σαφές. Ε, ε, μία μεγαβατόρα επί 10 ε, στη 12η ε, είναι μια τεραβατόρα. Ολοκληρώθηκε έτσι η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10 η ώρα για τις ψηφοφορίες σας. Παρακαλώ φέρτε μαζί σας τις κάρτες ψηφοφορίας σας οι συντονιστές θα συναντηθούν στις 9 η ώρα. Διακοπή της συνεδρίασης. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους. I don't. I don't like voluntary agreements either. I I won't say who's responsible for that inside the Commission.